So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τη συνεδρίασή μα. Ε, καλωσορίζω λοιπόν θερμά τον ε, Πρωθυπουργό του Συμβουλίου και Υπουργό Γεωργία τη Σουηδία, ε, τον κύριο Έσκιλ Έλαντσον. Καλώ ήρθατε κύριε Έλαντσον στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε πολλά κοινά σημεία μεταξύ των ε, θεμάτων ε, που επιλαμβάνεται η παρούσα Επιτροπή και της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Προφανώς και είναι πολύ σημαντική η συμβολή της γεωργίας στα περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα στο ζήτημα των κλιματικών μεταβολών και καθώς είμαστε και αρμόδια επιτροπή για την ασφάλεια των τροφίμων έχουμε να κάνουμε και με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Γνωρίζουμε πως ε, η Σουηδική Προεδρία ε, έχει θέσει υψηλούς στόχους στον εαυτό της, είναι ιδιαίτερα ενεργή και γνωρίζουμε πως έχει διαμορφώσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, οπότε θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα μας πείτε. Έχετε το λόγο κύριε Λαντσόν και πάλι καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ και με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας στον χώρο της Γεωργίας και της Αλληλείας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας να ξεκινούμε την Προεδρία μας ενώπιον ενός τόσο νέου, εκλογέτους δηλαδή, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, και θέλω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τα όσα θα μου δώσετε εσείς ως δικές σας απόψεις, ως δικό σας μήνυμα σε μένα ως ε, Υπουργό Γεωργίας αλλά και ως ε, Πρόεδρο του Συμβουλίου. Έχω υπάρξει για μεγάλη, μεγάλη διάρκεια των βουλευτή στο Συνδικό Κοινοβούλιο και γνωρίζω πώς αισθάνεται κανείς όταν βρίσκεται στην αρχή της βουλευτικής του θητείας και ε, πραγματικά θεωρώ πως ε, θα λάβουμε έτσι μια ενίσχυση ε, από σας με αυτή τη συζήτηση που θα γίνει. Υπάρχουν ούτως ή άλλως μια σειρά από τομείς αρμοδιότητες οι οποίοι είναι εκείνοι για το δικό μου Υπουργείο και για την Επιτροπή αυτή. Και ούτως ή άλλως οι περισσότεροι Υπουργοί θα έρθουν και θα μιλήσουν στη δική σας ε, επιτροπή. Για παράδειγμα το πρωί γνωρίζω πως είναι το συνάδελφός μου ο κύριος ε, Κάλγκρεν, ενώ αύριο θα παρευρεθούν εδώ στην επιτροπή σας ε, ο Υπουργός Κοινωνικής ο Γκέραν Χάγκλουν και η Μαρία Λάσσον, Υπουργός της Ηλικίας Δημόσιας Υγείας. Εμείς τώρα έχουμε τρία, τρεις ε, τομείς οι οποίοι από τις δικές μου αρμοδιότητες και οι τρεις βασίζονται στην χρήση χωρίς κατάχρηση ε, αλεία και κλιματικές μεταβολές και ταυτόχρονα υγιής, χρηστή, κτηνοτροφία. Και προφανώ και αυτά τα ζητήματα από τις δικές σα αρμοδιότητα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των κλιματικών μεταβολών, προφανώ εδώ έχουμε τι μεγαλύτερε ε, προκλήσει. Ολόκληρη η Ευρώπη αλλά και ολόκληρο ο κόσμο ε, δραστηριοποιείται αυτό το φθινόπερο σε αυτό το τομέα πάρα πολύ, καθώ ε, η Γεωργία παίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά το φαινόμενο των κλιματικών μεταβολών. Και θα πρέπει να σκεφτούμε το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων, ε, τις νέες ε, νόσους ε, τόσο φυτών όσο και ζωονόσους. Άρα λοιπόν εδώ εμπλέκονται όλα αυτοί οι τομείς όπως και ο τομέας της χρηστής ε, παραγωγής ενέργειας και διαχείριση της ενέργειας. Και μάλιστα είχαμε ε, μία συνεδρία του Συμβουλίου με βάση το κείμενο της Επιτροπής ε, με θέμα την συμβολή της γεωργίας στην, στις κλιματικές μεταβολές και η συζήτηση που θα γίνει στο Βέξο, στο θα εστιάσει και πάλι στις κλιματικές μεταβολές και συγκεκριμένα στο πώ μπορούν να μειωθούν οι εκπομπέ θεαριών του θερμοκηπίου από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Γεωργίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι κλιματικέ μεταβολέ, θα έχουμε δύο ακόμα συνεδριάσεις στη Σουηδία. Η πρώτη από αυτέ θα είναι ε, η σωστή διατροφή σε σχέση με την ενέργεια, ε, δηλαδή το πώ μπορούν οι καταναλωτέ να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε αυτό το τομέα καθώ το επιθυμούν. Και η δεύτερη διάσκεψη θα αφορά τον τομέα τη έρευνα. και συγκεκριμένα τις ε, αγροτικές περιοχές ε, και το πόσο μπορούν αυτές να συμβάνουν στη καλύτερη διαχείριση των κλιματικών μεταβολών. Εδώ ε, αναφερόμαστε ειδικότερα στο ζήτημα της βιώσιμης παραγωγής βιοενέργειας. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διάσκεψη που θα λάβει χώρα τέλη Σεπτεμβρίου με θέμα νερό και ε, Γεωργία, γιατί προφανώς η ποσοτική διαχείριση του νερού στη Γεωργία αποτελεί ένα κέριο ζήτημα για πολλά κράτη-μέλη. Ελπίζουμε λοιπόν πως εκεί ε, ε, στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων θα γίνουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Από εκεί και μετά έχουμε και το FLEGT, δηλαδή το FLEGT, και την ενίσχυση, περαιτέρω ενίσχυση της δασοκομίας. Εδώ έχουμε μία πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένε διατάξεις σε ό,τι αφορά τον χώρο τη υλοτομία και των όσων δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Ε, μιλάμε εδώ για ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο ε, και για ένα κείμενο το οποίο αφορά σε περισσότερους από ένα τομείς. Ε, το Συμβούλιο έχει ήδη δραστηριοποιηθεί εδώ και εσείς ως ε, Κοινοβούλιο. Την Άνοιξη μάλιστα εφετήσατε τη δική σας άποψη και προβήκατε σε κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα πρέπει ακόμα να αναλυθούν. Κατά τελευταία προεδρία εστιάστηκαν οι προσπάθειες στην επίτευξη μιας συνένεσης, μιας συμφωνίας έως τον Ιούνιο, αλλά ε, καθώς ε, υπήρξαν περαιτέρω συζητήσει στο επίπεδο του Συμβουλίου, δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία, οπότε αυτή είναι η προτεραιότητά μας, δηλαδή τέλη του φθινοπόρου να φτάσουμε σε μια συμφωνία στο Συμβούλιο. Τρίτη προτεραιότητα τώρα, στην οποία αναφέρθηκα, είναι η, η σωστή, η χρηστή κτηνοτροφία και ευημερία των ζώων. Δηλαδή θεωρούμε πως η σωστή κοινοτροφία αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία των ζώων και ταυτόχρονα για την εμπιστοσύνη ε, των καταναλωτών στο χώρο της κοινοτροφίας. Θα γίνει τον Οκτώβριο, θα λάβει η χώρα μια σχετική διάσκεψη και ελπίζω εδώ πως θα, θα υπάρξει ενεργός ε, ε, συμμετοχή και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια υγιή κοινοτροφία. Ε, σε σχέση με την ευημερία των ζώων, πράγμα το οποίο βέβαια θα συζητηθεί μετά και στο επίπεδο του Συμβουλίου. Υπάρχουν ε, διατάξεις, ε, μέτρα για την προστασία των ζώων που έχουν τεθεί επιτάπητος και για παράδειγμα ως προς το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν γενικά τα ζώα στον επιστημονικό τομέα. Επίσης υπάρχει και ένα κοινό σχέδιο σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων και με αυτό το ε, θα Σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων θα ήθελα να αναφερθώ εδώ με έμφαση στην, ε, στο έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία των ζώων θα υπάρξει μια αντίστοιχη νομοθετική πρόταση που θα βασιστεί σε αυτό το έγγραφο και η οποία θα υποβληθεί αρχές του 2010. Προφανώς ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές ώστε να ανταποκρινόμαστε στο σημερινό τρόπο εκτροφής των ζώων αλλά ε, προκειμένου και για να ε, ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι για την υγεία τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων Ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποιε βελτιώσει, ώστε ε, να είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των διατάξεων δηλαδή ούτω ώστε αυτές να είναι και πιο αποτελεσματικέ και να μην δημιουργούν ε, περιττή γραφειοκρατία. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα των τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων προφανώ είναι ένα ζήτημα το οποίο μα απασχολεί όλου, καθώ είμαστε όλοι καταναλωτές. Δηλαδή θέλουμε να γνωρίζουμε κατά πόσο τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε οι ίδιοι και τα παιδιά μα είναι θρεπτικά είναι υγεία αλλά ταυτόχρονα είναι και ασφαλή. Ειδικότερα σε αυτό λοιπόν το τομέα ε, των τροφίμων ε, είναι ε, πολύ σημαντικό το να υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις ειδικότερα για τον κλάδο. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στα νέα είδη τροφίμων, novel food και ταυτόχρονα στην ενημέρωση των ε, καταναλωτών, στην πρόταση δηλαδή την σχετική σε ό,τι αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη σχετική ενημέρωση. Σε ό,τι αφορά τα νέα είδη λοιπόν τροφίμων, των novel food, ε, να πούμε ότι ε, η σχετική ε, το σχετικό έγγραφο θα υιοθετηθεί από την πλευρά του Συμβουλίου μέσα στι ερχόμενε εβδομάδε και θα περάσουμε μετά στη δεύτερη ανάγνωση. Είναι φιλόδοξο αυτό, αλλά πραγματικά θα επιμείνουμε και θέλουμε να συζητήσουμε με τους, και να συνεργαστούμε πολύ στενά με τους αισιόδες συζητητές και με την Επιτροπή του ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το ταχύτερο δυνατό μία αποδεκτή λύση, ένα αποδεκτό συμβασμό και θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να ε, χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Χρειαζόμαστε πραγματικά πολύ μοντέρνα, πολύ σύγχρονη νομοθεσία ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις σημερινές συνθήκες και θα να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις για, μια καινοτόμο, για ένα καινοτόμο κλάδο ε, τροφίμων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έγγραφο, σε ό,τι αφορά τη διάθεση στην αγορά. Αυτό έλαβε πολύ δημοσιότητα και θα πρέπει να φτάσουμε στο σωστό ισοζύγιο, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε συνειδητή επιλογή ο καταναλωτή χωρί ταυτόχρονα να προβλέπουμε υπερβολικά πολλέ επιβαρύνσει για τον ε, παραγωγό. Ε, έχουμε ασχοληθεί πολύ εντατικά και εμεί και εσεί στο Κοινοβούλιο με αυτό το ζήτημα, αλλά ε, καλύπτει διάφορου τομεί και στο Συμβούλιο υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, οπότε βρίσκουμε μάλλον απίθανο το να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία μέσα στο φθινόπωρο. Εμεί ω Ιουδική Προεδρία ε, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε, να, να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια συνένεση μέχρι δηλαδή τα τέλη του έτους και της θητείας μας. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στα παραστοκτόνα. Ε, και εδώ έγιναν πολλοί εντατικέ διαβουλεύσει και διαπραγματεύσει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και καταφέραμε να ε, φτάσουμε σε μια συμβιβαστική λύση για τα τρία σχετικά νομοθετήματα. Όμω η τελευταία συνένεση που επιτεύχθηκε δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στην πράξη. Ε, αναφέρομαι συγκεκριμένα στα στατιστικά δεδομένα. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από την πλευρά της ε, Σουηδία είναι να φτάσουμε σε μια απλή και αποδεκτή λύση ώστε τελικά η συνένεση να επιτευχθεί, επιτευχθεί στη δεύτερη ανάγνωση. Αυτά λοιπόν ενημερωτικά κυρίε και κύριοι συνάδελφοι ω προ τα όσα θέλουμε να κάνουμε, ω προ του στόχου που έχουμε και βέβαια αναμένω τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον να μου πείτε ε, όσα θέλετε να μου πείτε για την ε, δική μα ε, Προεδρία κάτω στου επόμενου μήνε. Ευχαριστώ τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Λαντσόν. Ε, Μα αναφερθήκατε εδώ σε ένα από την πουρήση μια σύνθεση από πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα θέματα. Περνάμε κατευθείαν λοιπόν ε, στο ψητό. Ο κύριο Πενταλίζη έχει το λόγο. Ε, κύριε Λίζε, διακόπτει ο πρόεδρο. Τρία λεπτά χρόνο αγόρευση για όλου. Ναι, θα είμαι ακόμα πιο σύντομο. Θα αναφερθώ στην ασφάλεια των τροφίμων, πρόεδρε. Ε, και ειδικότερα στο ζήτημα του novel food, των νέων ε, τροφίμων, στο οποίο αναφερθήκατε. Γνωρίζετε πως ε, υπήρξαν εντατικές διαβουλεύσεις εδώ στο Κοινοβούλιο και πως η πολιτική συνένεση δημιούργησε κάποιες δυσκολίες και οδήγησε και σε μεγάλη συζήτηση και στο και, και έλαβε και μεγάλη δημοσιότητα, δηλαδή το κρέας από κλωνοποιημένα ζώα. Ε, το Συμβούλιο είπε πω ε, θα πρέπει να κινηθούμε βασικό προσανατολισμό την απόλυτη απαγόρευση και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει και μελλοντικά. Ε, και βέβαια θα πρέπει να μα απασχολήσει και η προστασία των ζώων σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή δεν έχουμε το να κάνουμε μόνο με την ασφάλεια, αλλά από την άλλη πλευρά είναι σαφέ ότι τα ζώα αυτά υποφέρουν. Άρα λοιπόν νομίζω πως και στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα πρέπει να θέσουμε τα και αυτό το επιχείρημα αν θέλουμε να προβούμε στη διακριτική μεταχείριση, δηλαδή να θέσουμε το επιχείρημα τη προστασία των ζώων. Άρα λοιπόν η πρόταση και η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο δεν μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αυτό να το πούμε. Μετά, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έπαιξε κάποιο ρόλο, ακόμα και κατά την προεκλογική περίοδο είναι τα προϊόντα απομιμήσεις, ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα είδη τυριού. Ε, μπορούμε να έχουμε εδώ κάποια ε, πρακτική σήμανση αυτών των προϊόντων τους ώστε να είναι πιο κατανοητή και για τους καταναλωτές από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Επίσης κάτι ακόμα θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την σήμανση των τροφίμων και το σχετικό κανονισμό. Είπαμε εμεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου ότι δεν θέλουμε να ασκήσουμε φοβερέ πιέσει, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Ε, καθώς είχαμε ε, και κάποιες ε, συζητήσεις που έγιναν επί μακρόν, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το αλάτι μέσα στο, στο ψωμί και ούτω καθεξής. Οπότε ε, ακόμα δεν ήμασταν σε θέση να επιτύχουμε μια πολιτική συνένεση. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ε, δεν αντιλήφθηκα στο τέλος της παρέμβασής σας όταν είπατε ότι η τελική ένεση ακόμα εκκρεμεί. Ελπίζω να αναφέρεστε σε τέτοιες ε, περιπτώσεις σε κείμενα τα οποία ήδη έχουν συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε πρώτη ανάγνωση. Αλλιώς ε, γνωρίζετε πως έχουμε ε, ποιες διαδικασίες ισχύουν. Δηλαδή ε, δεν μπορεί να υπάρξει μια οριστικοποίηση της θέσης ε, εάν δεν έχει επέλθει μια συζήτηση καταρχήν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλους τους στόχους που έχετε θέσει, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη αλληλεία. Ε, θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά ε, με τα συνολικά επιτρεπόμενα λιεύματα, με το μέγεθος του, ε, το, ματιού των δικτυών και ούτω καθεξής καλώς, αλλά μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ και άλλα ζητήματα ε, τις δηλαδή και την, ε, τις τους στα, στα ψάρια ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Βαλτική Έχουμε λοιπόν αυτά τα είδη ψαριών τα οποία συχνά τελικά καταλήγουν να γίνονται ζωοτροφές αλλά τελικά με αυτόν τον τρόπο ε, τέτοιου είδου ε, διοξίνες ε, ξαναμπαίνουν στην τροφική αλυσίδα οπότε έχουμε επανειλημμένα προτείνει στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα την υγιή, τη χρηστή κτηνοτροφία είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος σας ε, και αξιέπαινος, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς εννοείτε εδώ. Τι θέλετε να κάνετε, δηλαδή να καταγράψετε το πώς ακριβώς λαμβάνει η χώρα η κτηνοτροφία, η εκτροφή των ζώων. Καλώς, εντάξει, αλλά έχουμε να κάνουμε και ε, ε, κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν, σας ζητώ να μου πείτε, ή τουλάχιστον να μου, να δώσετε μια διαβεβαίωση ότι οι χθιάλευρα δεν θα αποτελέσουν ζωοτροφές για μερικαστικά γιατί αυτό το πρόβλημα έχει ε, ε, προκύψει ε, ξανά και ξανά. Δηλαδή τουλάχιστον μετά από την πρώτη φάση της ηλικία όταν έχει δηλαδή διαμορφωθεί πλέον το στομάχι αυτών των μερικαστικών, να μην τρέφονται σε καμία περίπτωση με ηχθιάδευρα. Επίσης, η εντατική και εκτατική γεωργία σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε ε, μικρότερους αριθμούς ζώων που θα εκτρέφονται στις ίδιες εκτάσεις, οπότε δηλαδή θέλουμε εδώ ένα μεγαλύτερο, ε, ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη διασπορά. Και επίσης κάτι ακόμα θα ήθελα να, να αναφέρω είναι η προστασία των ζώων. Εάν θα ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να υπάρξει μια ε, μεγαλύτερη πρωτοβουλία από την Πράξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι διάφορε επιτροπέ σε ό,τι αφορά το κυνήγι τη φάλαινας αλλά και τη φόκια. Ε, ούτως ώστε πραγματικά εκεί, στο πλαίσιο αυτών των επιτροπών, να λαμβάνονται ε, υπόψη και οι στόχοι της βιωσιμότητας. Ε, γιατί δεν είμαι βέβαια ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κυνήγι της φαλενάς. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις στον ΠΟΕ, ο κ. Λίζα αναφέρθηκε στο ζήτημα του κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα και εδώ το καταστατικό λέει ότι ένα κράτος μπορεί για λόγου, ηθικούς, για παράδειγμα για λόγου προστασίας των ζώων, να δημιουργήσει ένα εμπόδιο, ένα ε, εμπορικό ε, ένα κόλλημα κατά το εμπόριο και ελπίζω να μπορέσει να αξιοποιήσει, αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη δυνατότητα γιατί νομίζω πως συμφωνούμε από αυτού όλοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη-μέλη. γιατί για παράδειγμα ήμασταν και εκείνοι που πρώτοι αξιοποιήσαμε αυτή τη ρήτρα στο πλαίσιο του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά την ε, χρήση του δέρματος από σκύλους και γάτες. Επίσης, ε, ε, για παράδειγμα, σε ό,τι ή μάλλον θα ήθελα να αναφερθώ και στο ζήτημα του κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κρέατος με ορμόνες. Παρότι έχουμε ήδη αποδείξει ότι τέτοιου είδους ε, κρέας μπορεί να οδηγήσει, ε, να είναι καρκινογόνο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ε, παρενέργειες και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει κάτι, αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο. Δηλαδή να πρέπει να καταβάλουμε σχετικές πληρωμές για κάθε είδους προϊόντα, ως αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να συνεχίσει κάτι τέτοιο με το κρέας από τη ΣΥΠΑ. Um, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Υπουργό και για την παρουσίασή του. Αναφερθήκατε στις υποχρεώσεις ε, ε, των παραγωγών ε, που προμηθεύουν την αγορά με ξυλία και προϊόντα ξυλίας. Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο ψήφισε ήδη από τον Απρίλιο για το κείμενο αυτό και υποτίθεται ότι έπρεπε να δώσουμε καιρό στο Συμβούλιο και ε, τουλάχιστον για μία πρώτη ανάγνωση ή τουλάχιστον να είχαμε μία ε, συμφωνία πριν από το καλοκαίρι. Όμως ε, δεν, υπάρχει, δεν υπήρξε καμία συμφωνία και δεν βλέπουμε το Συμβούλιο να βιάζεται. Θα ήθελα να μας καθησυχάσετε και να μας πείτε ότι όντως θεωρείτε ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και για σας και ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Επίσης, εμείς θέλουμε να υπάρξει μία πλήρης απαγόρευση της, παρα... της θέσης σε... στην αγορά της παράνομης ξυλίας. Εμείς θέλουμε βέβαια να έχουμε μία φιλόδοξη συμφωνία, διότι στον δρόμο προς την Κοπενχάγη η αξιοπιστία μας ε, θα διακυβευτεί. Εάν δηλαδή δεν μπορούμε να, καθορίσουμε, να, να, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να καθαρίσουμε την αγορά μας από την παράνομη ξυλία... Ε, και ζητάμε μια πρόταση της Κομισιόν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, η Κομισιόν τελικά την υπέβαλε, αλλά έχει, βρίσκεται η πρόταση αυτή στο σιρτάρι του Συμβουλίου. Λοιπόν, επειδή πριν από την Κοπενχάγη πρέπει να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας, θα ήθελα πριν τουλάχιστον από τα Χριστούγεννα να υπάρξει μια συμφωνία. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό που ήρθε σήμερα εδώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η γεωργία και το περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και είναι σημαντικό να, ληφθεί, να λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο αυτής της αλληλεξάρτησης. Κάποια πράγματα θα ήθελα να τονίσω όμως. Το ένα είναι ότι θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι κάποια πράγματα δεν θα εμφανιστούν ξανά κατά τη διάρκεια της Σουηδικής ε, ε, Προεδρίας. Δεύτερον, ε, η αλλαγή για την αλλαγή του κλίματος, ότι θα το λάβουμε αυτό υπόψη μας και για την γεωργία. Και λαμβάνοντας υπόψη τώρα της, ε, την υιοθέτηση κανονισμών θα πρέπει να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση ε, όσον αφορά τον σεβασμό στις ε, τοπικές παραδόσεις κυρίως όσον αφορά τις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και την κτηνοτροφία και πώς επηρεάζουν όλα αυτά το περιβάλλον. Υπάρχουν σημαντικές επιστημονικές έρευνες ε, για τον περιορισμό της, ε, των εκπομπών αερίων ε, των, από τα ζώα, με, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διατροφή. Τρίτον, για την βιοπικιλότητα, οι αλλαγές στην, της, γεωργικής, της πολιτικής επηρεάζουν τη διοπικιλότητα, τα διάφορα είδη, ε, λαμβάνοντας τα πουλιά υπόψη σε συγκεκριμένο παράδειγμα, πολλές φορές δείχνουν την, τα καλά και τα κακά της εφαρμογής της γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα, μια ύπεθρο η οποία να είναι πιο φιλική προς τα πουλιά, αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι η εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής επηρεάζει την βιοπικιλότητα και την ε, ε, υγεία των πουλιών. Λοιπόν, θα, ε, αυτό το οποίο θέλαμε να, ζητήσουμε είναι, επειδή θα γίνει ούτως ή άλλως η αλλαγή του κλίματος, να προσαρμοστούμε όσο να τον περισσότερο και καλύτερα. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ ζητώ συγγνώμη, έπρεπε καταρχήν να βρω ένα μικρόφωνο. Εγώ είμαι η συγκήτρια σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη σήμανση ζωοτροφίμων και δεν ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε αυτό το ζήτημα βασικά γιατί ε, η Σουηδική Προεδρία δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το ζήτημα. Ε, η Επιτροπή είχε αποφασίσει κατά, τελευταία, ε, κατά το τέλος της βουλευτικής θητείας ε, να αναβάλει την πρώτη ανάγνωση ε, για, την ε, επόμενο, για το επόμενο κοινοβούλιο, δηλαδή για τη νέα κοινοβουλευτική θητεία, καθώ είχαν υποβληθεί πάρα μα πάρα πολλέ τροπολογίε, πράγμα που καταδεικνύει το ενδιαφέρον. Όμω, καθώ αναφέρθηκε ο συντονιστή, ο κ. Πέτα Λίζε, σε αυτό το ζήτημα και στο ζήτημα και της, των παραποιημένων προϊόντων, ε, πράγμα το οποίο φυσικά έχει να κάνει και αυτό με τη σήμανση των τροφίμων, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχει αναλογιστεί αυτά τα ζητήματα το Συμβούλιο ε, συνολικά, αλλά θα ήθελα να θέσω και το εξή ερώτημα. Ε, το δηλαδή προεκλογική περίοδο μετά διακοπές διακόπηκαν οι εργασίες του για το καλοκαίρι ενώ εσείς συνεχίζετε να εργάζεστε θεωρείτε πως ε, έχουν επιτευχθεί κάποια βήματα εδώ. Ε, έχει αναμείνει το Κοινοβούλιο ή έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μία άποψη από την πλευρά του Συμβουλίου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας να το ξέρουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε σήμερα μαζί μας και συζητείτε όλα αυτά τόσο σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι είναι ευτυχές το ότι προσπαθείτε να διασυνδέσετε τις καλές πρακτικές μερίες των ζώων, την καλή ποιότητα της κτηνοτροφίας για τα ανθρώπινα. Αυτό νομίζω είναι κάτι το πολύ θετικό. Επίσης, ένα άλλο θέμα μας απασχολεί, το θέμα της χρήσης αντιβιωτικών. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες ουσίες οι οποίες υπάρχουν ακόμη και στις ζωοτροφές αντιβιωτικές, αλλά βλέπουμε να υπάρχει ίσως και αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Πολλές φορές ε, συνταγογραφούνται και αντιβιωτικά ακόμη για τα υγιή ζώα. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει ώστε να μην αρχίσουν να παρουσιάζονται και στα ζώα βακτηρίδια πολύ ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δείτε στα πλαίσια της δική σας προεδρίας τι γίνεται στην κτηνοτροφία και πώς μπορούμε να έχουμε υγιή ζώα. Καθώς και να κάνουμε και στατιστικές για να δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά και να θέσουμε ενδεχομένως κάποιους στόχους μείωσης της χρήσης τους. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφορετικά, κάποια στιγμή δεν θα έχουμε πλέον φάρμακα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κάποια νοσήματα ακόμη και βασικά. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχετε να απαντήσετε σε πολλά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ για την ε, συνεισφορά σας και τις παρεμβάσεις που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εύστοχες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα αρχίσω πρώτα απ' με το novel food. Όντως, πρόκειται για ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα και είμαι πεπισμένος ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, υλοποιήσουμε αυτή τη ε, συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μια σύγχρονη νομοθεσία που να μας επιτρέπει να έχουμε ασφαλή διατροφής για τον άνθρωπο. Θα πρέπει να ξέρουμε βεβαίως ότι τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα. Σε θέματα ειδών διατροφής ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες και πακέτα νομοθετικών πράξεων αρκετά πολύπλοκα. Και υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν, κυρίως να μην ξεχνούμε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται η αρχή της ε, προσοχής για κάποια θέματα. Το... Για το τυρί φερρυπίν, που είναι ένα ευαίσθητο προϊόν. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε εάν θέλουμε να φτιάξουμε τυρί. Γάλα, κατά βάση, και σχεδόν τίποτε άλλο. Μπορούν να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, και προσωπικά πρέπει να πω ότι με λύπη μου διαπιστώνω να υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτό το θέμα, εξαιρέσει στους κοινοτικούς κανόνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού οι εξαιρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει το βασικό για μένα είναι και ο βασικός κανόνας, ο γενικός κανόνας είναι ότι για να φτιάξουμε τυρί πρέπει να έχουμε γάλα. Όλα τα άλλα θα πρέπει να είναι μικροεξαιρέσεις. Τόσο όσον αφορά τα παστοκτόνα, Πιστεύω ότι υπάρχει σε σχέση με τις στατιστικές μια κάποια παρανόηση. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες και αποκλίνουσες απόψεις για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όσον αφορά την αλία, πρόκειται για μία από τις πολιτικές προτεραιότητες ε, για την Σουηδική Προεδρία και γνωρίζουμε ότι αυτή η πολιτική έχει και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν την αλία. Η ποιότητα των υδάτων και θα πρέπει να ενεργούμε με τρόπο ώστε και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, καθαρά ύδατα για να ψαρεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι έχει κάνει μια κάποια πρόοδο και ξέρουμε ότι έχουν ε, εγκριθεί και κάποια διοικητικά σχέδια για να μπορέσουν να αποκατασταθούν τα αλλιευτικά αποθέματα. Δεδομένου ότι ξέρουμε ότι κάποια είδη είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Βλέπουμε λοιπόν να έχει αντιστραφεί σήμερα η τάση αυτή και βλέπουμε όλα σχεδόν τα θαλάσσια είδη να υπάρχουν στους πάγκους των σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία σωστή διατροφική αλυσίδα. Επίσης, οι απορρίψεις διοξίνης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε για να μην υπάρχουν κατάλοιπα στα είδη διατροφής που καταναλώνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της διατροφικής αλυσίδας. Κάποια άλλη ομάδα ερωτήσεων αφορά τα θέματα βελτίστων πρακτικών για την κτηνοτροφία και τα υγιή ζώα. Ζώα τα οποία ζουν σε καλές συνθήκες είναι ευτυχισμένα ζώα. Που παράγουν τα είδη διατροφής που χρειαζόμαστε υπό καλές συνθήκες. Ένα ζώο το οποίο δεν ζει σε καλές συνθήκες δεν μπορεί να είναι υγιές. Και γι' αυτό το λόγο προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις καλές πρακτικές για την κτηνοτροφία. Και φτάνω σε ένα από τα τελευταία ερωτήματα που τέθηκαν. Θέλουμε εμείς να μειώσουμε την χρήση αντιβιωτικών. Αν έχετε ζώα τα οποία ζουν σε καλές συνθήκες, αν έχετε υγιή ζώα, δεν χρειάζεστε αντιβιωτικά. Επαναλαμβάνω, εάν θέλουμε να μειώσουμε την χρήση αντιβιωτικών, θα πρέπει να έχουμε ζώα τα οποία να ζουν σε καλές συνθήκες στα πλαίσια των, ε, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τις οποίες μεγαλώνουν. Και θα ήθελα τώρα να επανέλθω στην ε, σημασία της αρχής προφύλαξης και να αναφερθώ και στο ε, θέμα στο θέμα το φυτογενομικό. Πρόκειται για μια αρχή την οποία θέλουμε να εφαρμοστεί δεδομένου ότι θεωρούμε ότι είναι σημαντική για τα είδη διατροφής. Είτε πρόκειται για είδη διατροφής για τον άνθρωπο είτε για ζωοτροφές. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο Flex. Πρέπει να νομοθετήσουμε για αυτό το θέμα με τρόπο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να έχουμε μία νομοθεσία που να αντιστοιχεί στις συμφωνίες που έχουμε συνάψει ανά τον κόσμο και σέβεται τις διάφορους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, να έχουμε ένα νομοθετικό πακέτο που να λαμβάνει υπόψη την ε, συμβατότητα με τις, ε, τους εμπορικούς κανόνες και ξέρουμε ότι η νομοθεσία την οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή αφορά πάρα πολλά άτομα και πάρα πολλούς τομείς. Τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς, τις τελωνιακές αρχές και λίγο όλους μας, δεδομένου ότι είμαστε όλοι καταναλωτές όταν πρόκειται για προϊόντα ξηρή, ξυλίας. Θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί αυτό το θέμα στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να επιτευχθεί η συμφωνία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία το Δεκέμβριο, αλλά δεν θα πρέπει να μακρηγορήσουμε και να περιμένουμε πάρα πολύ πριν να καταλήξουν οι συμφωνίες στο θέμα αυτό. Και ακόμη μια συμπληρωματική παρατήρηση αναφορά αφορά τα αντιβιωτικά. Όταν μιλούμε για νομοθεσία, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή η νομοθεσία γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν είναι σημαντική μόνο η εθνική νομοθεσία. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για όλους, και θα λάβω υπόψη αυτά τα οποία είπατε. Θα συζητήσω με την συνάδελφο Μαρία Λάρσεν που θα σας επισκεφθεί αύριο και θα προσπαθήσω να δω μαζί της πώς μπορούμε να διαθετήσουμε, να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό των αντιβιωτικών και πώς θα μπορέσουμε επίσης να το συζητήσουμε και να φράσουμε την άποψή μας και σε επίπεδο Σουηδικής κυβέρνησης. Έχω την φιλοδοξία σήμερα το απόγευμα να μιλήσουν όλοι. Είναι δέκα αυτοί που έχουν, είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλος. Λοιπόν, δύο λεπτά οι περισσότεροι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τις απαντήσεις που δώσατε στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτό που αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίες... τον τρόπο δηλαδή που θα διευκολύνεται τον μια βιώσιμη αλία. Πιστεύω ότι η θέση που αφορά τις ε, ποσοστώσεις στην αλία θα παίξουν, ε, ζωτική, θα παίξουν ε, μεγάλο ρόλο. αν διαβάσω σωστά εδώ το πρόγραμμα εργασίας σας και τις φιλοδοξίες που κρύβονται πίσω από αυτό ε, είναι σαν να θέλετε να πείσετε το Συμβούλιο οι, οι ποσοστώσεις να ορίζονται με βάση την, τις, ε, τα ψάρια. Ε, άρα τα, τα, τα, οι, οι ποσότητες των ψαριών θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο από τις οικονομικές συνέπειες όσον αφορά τον καθορισμό της, ε, των ποσοστώσεων. Η επόμενη ομιλήτρια. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να μου πείτε αν κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας θα συζητήσουμε και για τα θέμα ε, των ε, μεταλλαγμένων. Υπάρχει βιολογική ε, υπάρχουν, υπάρχει βιολογική καλλιέργεια, μετά μιλάμε και για τα ευτυχισμένα ζώα και εδώ κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για τους νέους τάβλους, πώς θα επιβάλλεται αυτή τη νέα μορφή των στάβλων σε όλη την Ευρώπη. Όταν μιλάμε για κλιματολογικές αλλαγές, πιστεύω ότι μιλάμε για λάθος, για λάθος πράγματα, με σε λάθος βάση. Υπάρχει το όζον, υπάρχουν οι πάγοι που λιώνουν, αλλά ε, οι συνέπειες ε, των κλιματολογικών αλλαγών θα έρθουν αργότερα. Τώρα όμως ε, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ο περιορισμός των πρώτων υλών. η βιομηχανική γεωργία δεν είναι βιώσιμη. Η Κίνα θα ε, απαγορεύσει την, ε, ε, τις εξαγωγές κάποιων πολιτήμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων. Όλη η αντιμετώπιση για την, για την πρόληψη της, των κλιματολογικών αλλαγών στηρίζονται σε λάθος βάση θα χάσουμε τους σπόρους μας, θα υπάρχει κατάρρευση ε, του περιβάλλοντος και θα υπάρξει ε, πείνα. Κυρίως όσον αφορά τα ορυκτά, το πετρέλαιο δηλαδή, ε, τα... Κάποιες, κάποια προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά για μας και σημαντικά για την, για την γεωργία μας. πιστεύω ότι δεν πρέπει να ε, χτίζουμε ε, παλάτια στην άμμο, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια είδαμε χαρά ότι αναφερθήκατε εκτεταμένα στην βιοπικιλότητα. Τα τελευταία χρόνια όμως η Νότια Ευρώπη πλήττεται συστηματικά από μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, χάνοντας περίπου 4 εκατομμύρια στρέμματα το χρόνο. Και η κλιματική αλλαγή, η οποία παρά την άποψη άλλων συναδέλφων έρχεται και την βιώσαμε εμείς στην Ελλάδα ήδη το 2007, με τις μεγάλες πυρκαγιές τότε, πρόκειται να επιδεινώσει τα πράγματα. Η δε Νότια Ευρώπη είναι κατεξοχήν ευάλωτη περιοχή, μας λένε όλες οι επιστημονικές μελέτες. Μία από τις πτυχές της επιδείνωσης είναι και η σοβαρή απώλεια βιοπικιλότητας, καθώς τα δάση αυτά χάνονται και δεν αναπαράγονται. Ε, προτίθεστε ως Προεδρία μέσα στα θέματα της βιοπικιλότητας να εξετάσετε και αυτό το πρόβλημα των δασών που καταστρέφονται στην Νότια Ευρώπη. Thanks very Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την παρουσίασή του και για τις απαντήσει που ήδη μα έδωσε. Θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο ζήτημα τη μα των ε, και στο οποίο αναφερθήκατε και ορθά είπατε ότι θα πρέπει να μπορούν ε, οι καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένη ε, επιλογή. Πράγματι θα πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία, ένα ισοζύγιο, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ισορροπία εδώ, εντός της ε, δικής μας Επιτροπής. Και ε, για να το κάνουμε αυτό ε, εν ώψη και τη ε, συζήτηση στην πρώτη ανάγνωση, θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στο ζήτημα τη χώρα προέλευση σε σχέση με τη σήμανση. Δηλαδή, λαμβάνω πολλέ αναφορές από ε, πολίτες ε, της δικής μου επικράτειας, ε, από Γεωργού σε ό,τι αφορά την, τις λανθασμένες αναφορές ως προς το από πού προέρχονται, ποια είναι η προέλευση δηλαδή των συγκεκριμένων προϊόντων. Θα θέλαμε να διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι είναι υποχρεωτική η αναφορά της χώρας προέλευσης, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα τρόφιμά τους, ειδικότερα για τα γαλακτοκομικά, για τα προϊόντα που αποτελούνται από μία από ένα κύριο συστατικό ε, και για τα κύρια τρόφιμα. Θα θέλαμε λοιπόν ε, να δούμε κατά πόσο ε, είσαστε διατεθειμένος να κάνετε κάτι ώστε να επιλύσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και να δείξετε αυτή την βούληση. Ναι, τα βρετανικά σούπερ μάρκετ θα σας πούνε ότι για παράδειγμα το λόγο προϊόν προέρχεται από την Ουαλία ή το άλλο προϊόν προέρχεται από την Σκοτία. Κυρία Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό που παρευρίσκεται σήμερα εδώ για να συζητήσει σήμερα μαζί μας τόσο από προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και από τη δική σας ε, κυβέρνηση της Σουηδίας ε, έχουμε ακούσει ε, πως η Βαλτική αποτελεί προτεραιότητα και ζήτημα μεγάλης σημασίας. Σας. αναφέρεστε στη Γεωργία, αλλά η Γεωργία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί ακριβώς το περιβαλλοντικό ζήτημα στη Βαλτική. Ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά τον αστροφισμό εκεί, αυτής της αυτό, αυτής της θάλασσας. Ε, ε, αυτός ο ευτρονισμός δημιουργείται κυρίως ακριβώς από ε, την γεωργία, από τα δικά της απόβλητα. Οπότε ενδεχομένως θα πρέπει κάποια στιγμή το Συμβουλίο να ασχοληθεί στα σοβαρά με αυτό το ζήτημα και σας ρωτώ. Πιστεύετε πως πραγματικά θα αλλάξει κάτι στις διατάξεις που προβλέπονται για τον χώρο της γεωργίας ώστε να μην καταλήγουν τόσα πολλά φωσφορικά άλατα και, και τόσο άζωτο στη Βαλτική. Ε, ε, ε, γίνονται κάποιες αναφορές οι οποίες όμως δεν είναι πολύ σαφείς σε ό,τι αφορά τα μέτρα δηλαδή που θα ληφθούν για την προστασία της Βαλτικής. Οπότε θα ήθελα και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, γιατί τελικά εσείς είσαστε ο Υπουργό Γεωργίας της Σουηδίας. Πείτε μας λοιπόν, έχετε προβλέψει συγκεκριμένε διατάξει οι οποίε θα οδηγήσουν πραγματικά σε βελτίωση τη περιβαλλοντική κατάσταση στη Βαλτική και μείωση των αποβλήτων φωσφορικών αδάτων και αζότου σε αυτή. Αν θέλετε κύριε Υπουργέ μπορείτε να απαντήσετε τώρα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω με τα θέματα της αλίας. έχουμε μία πρόταση για κάποια μέτρα τα οποία θα παρουσιαστούν σαν πακέτο και ελπίζω ότι θα υιοθετηθούν έτσι το φθινόπωρο διότι όταν μιλάμε για την αλία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όσον αφορά τις ποσοστώσεις. Διότι αν τα κράτη-μέλη καταλήξουν ε, σε κάποιες συμφωνίες για κάποια είδη, εάν αποφασίσουμε ας πούμε, ότι κάποιες ποσότητες ε, ψαριών δεν μπορούν να αλλιευθούν, τότε αυτή είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το λάβουμε υπόψη μας και στις προτάσεις ε, που υποβάλλουμε. Δηλαδή, όλοι πρέπει να σεβαστούμε τις ηλιμένες αποφάσεις. Και αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να ελέγχουμε και το τι γίνεται. Αυτό είναι βασικό. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την αρχή. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει και ένα σύστημα αποτελεσματικό ελέγχου, έτσι ώστε να εφαρμόζεται η κοινή αλληλευτική πολιτική από όλους. Επίσης, θα ήθελα να επαναλάβω κάποια πράγματα τα οποία ήδη έχουν λεχθεί. Μιλήσαμε πολλές φορές για ένα όραμα και όντως αυτό το όραμα είναι σημαντικό και εφαρμόζεται και στην αλία. Αλλά για να, μπορέσει, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αλία πρέπει να υπάρχουν ψάρια. Τα ψάρια δεν κατασκευάζονται από μηχανήματα, πρέπει να υπάρχουν στην θάλασσα. Άρα πρέπει να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία να μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την, τα ψάρια αυτά και να, να εξασφαλίσουμε την αναπαραγωγή τους. Και τώρα, τώρα το, το φθινόπωρο, θα υιοθετήσουμε κάποια μέτρα ελέγχου έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι σέβονται τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζονται οι... τα είδη των ψαριών στις διάφορες θάλασσες. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποιες, ε, κάποιες μεθόδους αλίες που δεν είναι τόσο επιλεκτικές. Εκεί ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχω επαναλάβει πολλές φορές μέχρι τώρα. Τώρα, για τους πόρους που μας προσφέρει η γη, όχι η θάλασσα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καλλιεργούμε χωρίς να καταστρέφουμε. Όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική ή για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα δάση, θα πρέπει να τονίζουμε ιδιαίτερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τρόπους και μεθόδους όπου θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Π.χ. ας πούμε στη Γεωργία, τα άχυρα. Πώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το, τα, τα βιοκαύσιμα. Σε αυτό τομέα αυτό κάποιες χώρες είναι πιο προχωρημένες από κάποιες άλλες και θα πρέπει να υποφεληθούμε από την εμπειρία κάποιων χωρών έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να ξεφορτωθούμε, αν θέλετε, να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας στο πετρέλαιο και στα άλλα ε, ορυκτά καύσιμα. Στην Σουηδία, ξέρετε, η Σουηδία είναι μια χώρα του βορρά, μια βιομηχανική χώρα που κάνει πολύ κρύο το χειμώνα και εκεί το 20% της ενέργειάς μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να τα καταφέρουμε αυτό, για να πετύχουμε αυτό το ποσοστό, το οποίο είναι αρκετά υψηλό ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιούμε κάθε ενδεχόμενο. Ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το χρησιμοποιούμε. Επίσης, η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Εφόσον υπάρχουν ε, πυρκαγιές ή εφόσον ε, υπάρχει μια φυσική καταστροφή ή υπάρχει διάβρωση του εδάφους ε, σε κάποιο κράτος μέλος, υπάρχει, ένα, υπάρχει αλληλεγγύη η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και να συνεργαζόμαστε μάλλον μεταξύ μας εφόσον υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Ήδη υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν και που και επιτρέπουν την αποδέσμευση κάποιων πόρων και την κατανομή τους σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, από την 1η Ιουλίου ήδη υπάρχουν δύο προγράμματα καταπολέμησης των πυρκαγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινωτικούς πόρους και κανονικά θα, μας, θα έπρεπε να, να μας επιτρέπουν την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα μπορούσα να προσθέσω ότι κάνουμε και κάποιους ε, ελέγχους, ε, κάποια health checks, ε, αν θέλετε, κάποιες, κάποιους ελέγχους που αφορούν την υγεία της γεωργικής πολιτικής και Ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, αποφασίσαμε να γίνει μια μεταφορά των πόρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε με τον τρόπο αυτό στη διάθεσή μας περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα της, των κλιματολογικών αλλαγών, της ε, έλλειψης ε, υδατίνων πόρων ή της αντιμετώπισης, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική για την Βαλτική, όντως ε, για μας τουλάχιστον, για τη Σουηδία, είναι ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας και αφορά όλη την Ευρώπη βέβαια και τις, τις όχι μονάχα τις χώρες που, είναι, που βρέχονται από την Βαλτική. Υπάρχουν πολλές... Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει το πρόβλημα των μεταφορών, υπάρχει το πρόβλημα των, ε, των, των αποβλήτων τα οποία ρίχνονται, χύνονται στην Βαλτική, υπάρχει το πρόβλημα της αλίας, της γεωργίας και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την Βαλτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και μία οδηγία για τα ζωτούχα, τα οποία επιτρέπουν τον, να, περιοριστούν οι συνέπειες της γεωργίας και μετά είχαμε, έχουμε και μία άλλη σειρά νομοθετικών κειμένων που επιτρέπουν την διατήρηση κάποιων ζωνών, κάποιων περιοχών όπου δεν χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα. Διατηρούνται καθαρές οι περιοχές αυτές. Πρόεδρε, νομίζω ότι απήντησα στις περισσότερες των ερωτήσεων που ετέθησαν. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε, έχουν στήσει άλλη συναδελφή το λόγο. Καταρχήν η κυρία Κριστίνα Τσιέρας Κορτίνης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Πρώτα απ' όλα, θα κάνω μία ερώτηση για να αναφέρω δύο θέματα τα οποία αναφέρετε εσείς. Το θέμα του ύδατος της γεωργίας και το θέμα των ζανιοκτώνων και φαστοκτώνων. Όλοι οι επιστήμονες που μελετούν το θέμα του ύδατος του κύκλου των βροχών και της κλιματικής αλλαγής συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε νομοθεσία με, χρησιμοποιώντας το ίδιο κριτήριο για τις χώρες του Ατλαντικού με τις χώρες της Μεσογείου. Διότι οι συνθήκες στις δύο αυτές ομάδες χωρών είναι εντελώς διαφορετικές και οι κλιματικές αλλαγές εντελώς αλλαγές. Το ίδιο σημαίνει και με τα ζυζανιοκτώνα και τα περιστοκτώνα. Η επιστημονική κοινότητα λοιπόν και η γεωργή των ε, νοτίων χωρών βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, δεδομένου ότι εφαρμόστηκαν για αυτούς κριτήρια που εφαρμόζονται στις χώρες του Βορρά και έτσι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Έτσι άνοιξε η αγορά για κάποια ζυζανιοκτώνα και ντομοκτώνα που προέρχονται από την Κίνα και που είναι κακής ποιότητας και βρέθηκαν στι αγορές μας. Γι' αυτό ε, ε, ρωτώ εγώ, πότε θα ασχοληθείτε αυτό, με αυτό το θέμα. Εάν καταλήγατε σε ένα μόνο συμπέρασμα μετά από την εξαμηνία ε, προεδρία σας, ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες χωρών και προσπαθούσατε και προσπαθήσετε να ενεργήσετε ανάλογα, θα ήμουν ικανοποιημένη. Πότε θα δούμε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, το θέμα της ασφάλειας των ειδών διατροφής. Η αρχή της αμοιβιότητας πότε θα εφαρμοστεί, διότι στις χώρες της Μεσογείου υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες περιορίζονται δεδομένου απαιτείται να χρησιμοποιούν ε, ειδικά ζυζανιοκτώνα, ενώ κάποιε επιχειρήσει ειδών διατροφή που βρίσκονται, κάποιες εταιρείε στις βορειοαφρικανικέ χώρες εισάγουν σε εμά ό,τι θέλουν και εδώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πότε λοιπόν θα ισχύσει αυτή η αρχή τη αμοιβαιότητα και πάλι, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπογραμμίσατε κύριε Υπουργή πόσο ε, σημαντικό θεωρείτε το να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά τις ε, βιολογικές καλλιέργειες. Ε, συγκεκριμένα θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι ακριβώς το ποσό, ποιο είναι το μέγεθος των κονδυλίων που θέλετε να διαθέσετε για την ενίσχυση της Πρόεδρος, ε, ο Κάρλ Σλίτερ ε, ως τελευταίος ε, ομιλητής. Εκτός και αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουν δύο ακόμα ή τρεις συνάδελφοι το λόγο. Καλώς. Κάρλ Σλίτερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην νανοσήμανση εμείς είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία στη σχετική έκθεση σε ό,τι αφορά την νανοτεχνολογία και από εκεί και μετά υπήρξε και έκθεση σε ό,τι αφορά τα νέα είδη τροφίμων, το Novel Food. Ε, αντίστοιχη συμφωνία υπήρξε ε, στο Συμβούλιο, οπότε θα ήθελα να ξέρω ε, τι συμβαίνει με τα νάνο σωματίδια και τα νάνο Έχει διαφοροποιήσει την άποψη του το Συμβούλιο ή εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά πάλι το ζήτημα των τροφίμων και την ασφαλεία τους, ε, ε, το Συμβούλιο είχε πει πω. Ε, ε, ε, θέλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της σήμανσης και των ζώων τα οποία έχουν λάβει ζωοτροφές από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Οπότε θα θέλαμε να γνωρίζουμε κατά πόσο πράγματι ισχύει αυτή η στάση του Συμβουλίου, ότι δηλαδή επιμένει σε αυτό στη σήμανση των σχετικών ζώων, γιατί βέβαια το ενόκο ζήτημα απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές μας. Θα κάνετε κάποια αντίστοιχα βήματα. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα που αφορά τις ε, νοροσυρά των Άλπαιων στη Γαλλία, όπου οι πρακτικές ε, κτηνοτροφίας και βοηδών σέβονται τη βιοπικιλότητα και τις παραδοσιακές μεθόδους. Δυστυχώς, οι κτηνοτρόφοι μας αυτοί έχουν όλο και περισσότερο ένα παραβανόμενο πρόβλημα, την παρουσία λύκων και την ε, συμβατότητα ή όχι αυτών με τα ε, ε, κτηνοτροφή αυτή καθεαυτή και με την προστασία αυτών των ζώων. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν κάποια συνοδευτικά μέτρα προστασίας των κτηνοτρόφων, διότι έχουν την εντύπωση ότι δεν ε, αναγνωρίζετε αυτή τη στιγμή πόσο σημαντική είναι η κτηνοτροφία ε, σε των βοηδών ε, στα ψηλά βουνά που σέβεται την βιοπικιλότητα και εξίσου πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστούν οι λύκοι που όλο και περισσότερο επιβιώνουν. Επίσης, θα ήθελα ένα άλλο πρόβλημα σημαντικό να αναφέρω. Η πτώση της τιμής του γάλατος για τους ε, γαλακτοκόμους. Αυτή τη στιγμή στην Γαλλία πολλοί γαλακτοκόμοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δίνη κατάσταση, διότι δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα που έκαναν και τις επενδύσεις που έκαναν για να σέβονται πραγματικά τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και να έχουν επεκτατική ε, κτηνοτροφία, και συγχρόνως δεν έχουν κανένα κέρδος. Θέλουμε να διασφαλιστεί η... ο κλάδος αυτός, θέλουμε να ανταποκρινόμεθα στα αιτήματα των καταναλωτών, να σεβόμεθα το περιβάλλον, να προστατεύσουμε και να διασφαλίσουμε την γεωργία και την γαλακτοκομία. Θέλουμε να μην εισάγουμε προϊόντα ε, αγροτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν μπορούμε εμείς να τα παράγουμε. Θέλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον. Έχετε λοιπόν εσείς, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα θέματα, ε, την πρόθεση να προτείνετε συγκεκριμένα μέτρα, δεδομένου ότι πρόκειται για επίγοντα μέτρα και συγχρόνως να προετοιμάσετε την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, η κυρία Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα τα οποία έχουν σχέση και με τις τελευταίες ερωτήσεις που έθεσε ο κ. Σίτερ για τις νανοτεχνολογίες. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό σήμερα κάποια είδη διατροφής να περιέχουν κάποιες νανοουσίες χωρίς να υπάρχει στην ε, ε, ετικέτα μια τέτοια ο κανονισμός Rich δεν αφορά τα ανανοσυστατικά. Σκέφτεστε να μελετήσετε το όλο το θέμα αυτό του καθεστώτος που θα διέπει τα ανανοσυστατικά. Ξέρουμε ότι στα καλλιντικά και στα είδη διατροφής έχουμε να κάνουμε με δύο θέματα πολύ σημαντικά για τον καταναλωτή. Και τώρα, μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ, σκέφτεστε κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας να μελετήσετε εκ βαθέων το είδος της γεωργίας που θέλουμε να έχουμε αύριο στην Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή ενθαρρύνουμε την γεωργική συγκέντρωση και τι λέμε, ότι θα θέλουμε να ε, έχουμε εντατική καλλιέργεια. Από την άλλη ενθαρρύνουμε τη χρησιμοποίηση των ε, παρασιτοκτόνων, αλλά θέλουμε να έχουμε μία σωστή καλλιέργεια και έχουμε υπερσυγκέντρωση αυτών των δραστηριοτήτων. Έχουμε πάρα πολλές καλλιεργούμενες γέες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται και όταν όλα είναι υπερσυγκεντρωμένα στη γεωργία πολλές φορές υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εξουδετέρωση όλες τις παραγωγές. Τι σκέφτεστε να κάνετε με όλα αυτά τα θέματα λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, ε, κύριο Υπουργό κατά πόσο οι εργασίες του κατά τη δική του Προεδρία θα συμπεριλάβουν τη σύνδεση ε, μεταξύ Γεωργίας και του Natura 2000 καθώς στη δική μου περιοχή υπάρχουν πολλές αντιθέσεις ε, μεταξύ του Natura 2000 και της Γεωργίας. Ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τον ε, κλάδο της Γεωργίας, ο οποίος έχει ψηλό κόστος από αυτήν την ιστορία. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος, η κυρία Μισελ Ερβάζη ως τελευταία ομιλητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε εδώ μαζί μας. Βλέπω ότι οι ερωτήσεις είναι παρόμοιες. Ε, στην Επιτροπή Γεωργίας η Επίτροπος Φίσερ Μπέλ είπε ότι το 80-90% της σόγιας που εισάγεται στην κοινότητα είναι μεταλλαγμένη. Γνωρίζοντας ότι την σόγια αυτή την δίνουμε, τη χρησιμοποιούμε για πρωτεΐνες στις ζωοτροφές, Πιστεύω ότι η σήμανση είναι ε, πάρα πολύ σημαντική για τους ε, καταναλωτές, ε, για να ξέρουν κατά πόσο καταναλώνουν μεταλλαγμένα προϊόντα ή όχι, και όσον αφορά το κρέας και όσον αφορά το γάλα. Επομένως, θα πρέπει στις, στην επισήμανση των προϊόντων θα πρέπει να, αναφέρεται η σόγια η οποία είναι μεταλλαγμένη. Τώρα, θα πρέπει να δούμε και τι είδους γεωργία θέλουμε διότι ούτως ή άλλως τώρα προωθούμε την ε, βιολογική καλλιέργεια. Λέμε ας πούμε ότι τα παιδιά μας και για την υγεία των παιδιών μας πρέπει να ε, ε, ε τους δίνουμε βιολογικά προϊόντα. Όμως είναι βιολογικά προϊόντα τα οποία ε, καλλιεργούνται στην Αργεντινή, καλλιεργούνται δεν ξέρω και εγώ πού, σε, ποια σημεία του πλανήτη και μεταφέρονται χιλιόμετρα ολόκληρα για να καταναλωθούν στην Ευρώπη. Επομένως είναι βιολογικά πετρελαϊκά προϊόντα θα έλεγα. Λοιπόν, πέραν όμως της βιολογικής ε, καλλιέργειας υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή να έχουμε λιγότερα ε, ζυζανιοκτώνα, λιγότερα πετρέλαια κτλ. Και ε, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι, πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουμε ε, έναν φόρο, ε, ε, φόρο άνθρακα για τα προϊόντα τα οποία διανύουν χιλιόμετρα ολόκληρα για να έρθουν να καταναλωθούν από τα παιδιά μας. Οι τελευταίες, αυτές είναι ο τελευταίες γύρες των ερωτήσεων. Η σειρά σας να απαντήσετε τώρα κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πολιτική των υδάτων και για τη σχετική οδηγία. Όλα τα και για τα παρασιτοκτόνα τα οποία χρησιμοποιούνται. Ξέρουμε ότι για το θέμα αυτό υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, περιφερειακές τοπικές πολιτικές και διαφορετικές προοπτικές. Όπως ξέρουμε, τα παρασιτοκτόνα διαλύονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το συστατικά του καθενός στα ευρωπαϊκά ύδατα. Προηγουμένως ξέχασα να απαντήσω σε κάποιο ερώτημα που αφορούσε την ε, σήμανση. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να πω το εξής. Όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτού για τα είδη διατροφής δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε συμπεράσματα. Υπάρχουν ακόμη προσυζήτηση κάποιες προτάσεις. Και για μένα θα πρέπει να υπάρχει σαφή σήμανση στα διάφορα προϊόντα για να ετημερώνεται ο καταναλωτής. Για να ξέρει τι ακριβώς αγοράζει. Επίσης είναι σημαντικό στην σήμανση να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να ξέρει ο καταναλωτής τι περιέχει το κάθε προϊόν και δεν θέλει εκείνος να καταναλώσει. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει ακόμη να αποσαφινιστούν για τις διάφορες ε, εταιρείες και θα πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για νέα νομοθεσία. Τώρα όσον αφορά την ε, δηλώσει για τον τόπο καταγωγής. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για τα είδη διατροφής. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις για το βόηο κρέας ή για τα νοπά προϊόντα. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι σημαντικό ο καταναλωτής να είναι πολύ σωστά ενημερωμένος. Όλοι στα σπίτια μας χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ε, προϊόντα τα οποία είναι σύνθετα ή που περιέχουν ε, συστατικά διαφορετικών τόπων καταγωγής, προέλευσης, αν θέλετε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν διάφορες αποκλίνουσες απόψεις στο Συμβούλιο. Θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να επιτύχουμε επαρκή πλειοψηφία για να καταλήξουμε στη συμφωνία. Όσον αφορά την ε, βιολογική καλλιέργεια, Έχουν δοθεί κάποια κονδύλια, έχουν μεταφερθεί κάποια κονδύλια από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη σωστά τα κονδύλια αυτά για να δουν τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια του πυλώνα 2 ώστε να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη ο καταναλωτής ε, στα διάφορα προϊόντα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, βιολογική καλλιέργεια. καλλιέργεια. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σχετικά κονδύλια για να ενισχυθεί η βιολογική καλλιέργεια. Μου κάνατε επίσης κάποιες ε, ερωτήσεις που αφορούν την ανατεχνολογία και τα ανανοσυστατικά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όντως πολλές φορές είναι δύσκολο να δούμε αν κάποια ε, είδη διατροφής είναι περισσότερο φάρμακα παρά είδη διατροφής. Για τα φάρμακα, τα κράτη-μέλη μπορούν πιο εύκολα ίσως να κανονίσουν τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να δουν κατά πόσον κάποιες ουσίες που θεωρούνται φαρμακευτικές ουσίες για μια χώρα δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά ειδών διατροφής από κάποια, άλλα, από κάποια άλλη. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη αρκετές δυσκολίες και είναι δύσκολο να δούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλούμε για σύνθετα προϊόντα ή για νανοτεχνολογίες. Τελειώνοντας, ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι που διαπιστώνω ότι όλα αυτά τα θέματα σας απασχολούν πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι όντως είναι δύσκολο να δοθεί προς το παρόν σαφής ορισμός στο θέμα των ε, νανοσυστατικών. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να καθορίσει προς το παρόν, αλλά είναι αυτό πολύ σημαντικό. Τώρα, για τις ε, γενετικά τροποποιημένες ουσίες και την ε, περιοκτικότητα κάποιων ειδών διατροφής σε τέτοιου ουσίες όσον αφορά και την μεταφορά κάποιων ειδών διατροφής. Θα ήθελα όλα αυτά τα θέματα να είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Σουηδική Προεδρία, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο, δεδομένου ότι περιμένουμε να υποβάλει πρόταση σχετικά με τα θέματα αυτά η Επιτροπή. Εάν όντω γίνει κάτι τέτοιο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια τη εξαμηνία Προεδρία μα. Αλλά ακόμη δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Όλα θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα με την οποία υποβάλει προτάσει η Επιτροπή. Και αν όντω υποβληθεί σχετική πρόταση, θα αποτελέσει αυτό το θέμα προτεραιότητα για μα. Τώρα, αφορά το γάλα και όλα τα θέματα που άπτονται της ε, λακτοκομίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι δυνατόν να κάνει μια ανάλυση της κατάστασης της αγοράς γάλακτος σε όλη την Ευρώπη. Η έκθεση της Επιτροπής την οποία ζήτησε το, ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπευλήθη 22 Ιουλίου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η αγορά γάλακτος στην Ευρώπη. Και το Συμβούλιο θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπόρεσε να γίνει η συνεδρίαση πριν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα και θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα με την έκθεση αυτή της Επιτροπής. Την έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνονται και διάφορες προτάσεις για την κατάσταση στην Ευρώπη και θα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό. Άρα προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο. Τελειώνοντας, για τις ζώνες Natura 2000 και το κόστος που απορρέει από την σχετική πρόταση, θα πω το εξής. Όπως ξέρετε, κάποια στοιχεία θα έπρεπε να μπορέσουν να ε, συμπεριληφθούν στον πυλώνα 2. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έκαναν διάφορες χώρες. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με δεχθήκατε σήμερα το απόγευμα και ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα είναι πολύ θετική κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας Σουηδική Προεδρίας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μια μεγάλη ποικιλία των θεμάτων την οποία θίξαμε, αλλά είδατε πόσο πολύ ενδιαφέρει τα μέλη της Επιτροπής μας σε ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό ήταν το κύριο ζήτημα, δηλαδή του να μην ε, έχουν τοξίνες, του να μην είναι επικίνδυνα τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Όλα αυτά λοιπόν μας απασχολούν. Ε, προφανώς και μας ενδιαφέρει και η συμβολή της ιεωργίας και της δασοκομείας στην ε, προστασία του περιβάλλοντος και ε, στην προστασία από τι κλιματικές μεταβολές και σε πολλά άλλα ζητήματα. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ελπίζουμε πως η συνεργασία μας θα είναι πολύ καλή. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τριών τεσσάρων λεπτών μέχρι να βρίσκεται εδώ μαζί μας ε, η κυρία Σουσάνα Γιάκομ από το ECDC για να προβούμε δηλαδή στην επόμενη συζήτηση. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Arbeit und es ist mir eine besondere Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επιστρέφουμε στι εργασίε μα και με μεγάλη μου χαρά ε, καλωσορίζω σήμερα ε, εδώ μαζί μα ε, την κυρία Σουζάνα Γιάκα, την Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Ε, σα ε, καλωσορίζω θερμά κυρία ε, Γιάκα, εδώ στην δική μα Επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου. Έχουμε μια σειρά από θέματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας και αναμένουμε βέβαια με ενδιαφέρον τα όσα θα μας ε, παρουσιάσετε τώρα σε σχέση με τις εργασίες σας και την οργάνωση της ε, δικής σας αρχής του δικού σας κέντρου. Και βέβαια μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ το ζήτημα της γρήπης ε, και εκεί θα θέλαμε βέβαια να ακούσουμε μεγάλο καλό πείτε. Έχετε λοιπόν το λόγο κυρία Ιακάπ, για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρο. Μέλη της ε, Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Είναι πραγματική τιμή για μένα που μπορώ να είμαι παρούσα σε μία από τις πρώτες συναντήσεις της Επιτροπής σας που δείχνει ότι, είσαστε, ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για το κέντρο και και όχι μόνο για και για τα θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολούμεθα. Ε, θεωρώ ότι η συνεργασία μαζί σας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχαμε και ένα επικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην προηγούμενη θητεία και πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή ήταν πολύτιμη για την δημιουργία και την λειτουργία στα πρώτα βήματα του, του, ε, ελπίζω ότι η σημερινή μας ε, συνάντηση θα καθορίσει το πρώτο βήμα ε, της νέας μας συνεργασίας με την, με την νέα Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να ξέρετε ότι όποτε με χρειαστείτε ή μας χρειαστείτε θα είμαστε στη διάθεσή σας. Εάν και εφόσον με χρειάζεστε ή έχετε κάποια θέματα στη μερική διάταξή σας που μας αφορούν, θα είμαστε εδώ. Και επίσης ε, θα καλωσορίσουμε στο ΕΚΠΕ ε, την αντιπροσωπεία του, ε, της Επιτροπής σας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας στέλνω συνέχεια επιστημονικά, επιστημονικές ενημερώσεις, αν θέλετε, για τις τελευταίες εξελίξεις. Και αν και εφόσον αποφασίσετε, κύριε Πρόεδρε, να δημιουργήσετε ένα σημείο επαφής αν θέλετε στην επιτροπή σας, ε, επαφής με το ΕΚΠΕ, ε, θα είναι ακόμα καλύτερα, όπως υπήρχε και στην προηγούμενη θητεία. Δεν θέλω να σας ε, φορτώσω με έγγραφα. Μπορώ να σας στείλω όλα τα έγγραφα, όλα τα έγγραφά μας, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω και να κατακλείσω, αν θέλετε, την επιτροπή σας. Θα μπορούμε να τα στείλουμε σε αυτό το σημείο επαφής και από εκεί και πέρα ανάλογα να διανέμονται. Το θέμα μας ε, είναι η πανδημία της γρήπης ε, ε, και θα αφιερώσω το δεύτερο κομμάτι της παρέμβασής μου σε αυτό το θέμα. Όμως πριν προχωρήσω στην θέμα της πανδημίας της γρήπης θα ήθελα να, παρουσ... να σας συστηθώ, να σας παρουσιάσω και, την... και τον οργανισμό μου όπως και το πρόγραμμα εργασίας μας. Το όνομά μου είναι Σουζάνα Γιάκαπ. Είμαι από την Ουγγαρία και είμαι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο ε, ε, Ασθενειών, το, ε, του ΕΚΠΕ δηλαδή, από τον καιρό που άρχισε να λειτουργεί το κέντρο το 2005. Πριν ήμουν υφυπουργό ε, υγείας ε, στην Ουγγαρία, Επίση εργάστηκα και στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία για 11 χρόνια σε, διάφορε διευθυντικέ θέσει. Όπω Όπως ξέρετε, η ΕΚΠΕ έχει την έδρα της, το ΕΚΠΕ μάλλον, έχει την έδρα του στη Στοκχόλμη και η, αποστολή του είναι να ενδυναμώσει τι την άμυνα της Ευρώπης απέναντι στις μολυσματικές νόσους. Ε, έχει έναν ρόλο σημαντικό στην αξιολόγηση, ε, αλλά και ε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να συμβουλεύουμε και να υποστηρίζουμε την Κομισιό με με επιστημονικά δεδομένα. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιό, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με, διάφορα άλλα, με διάφορους άλλους οργανισμούς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προφανώς. Τα τελευταία 4,5 χρόνια το ΕΚΠΕ από ένα άτομο το οποίο απασχολούσε, εμένα δηλαδή, και, με έναν, ε, και από έναν ετήσιο προπολογισμό κάτω από 5 εκατομμύρια, φτάσαμε σε, ένα, σε έναν οργανισμό που απασχολεί 250 άτομα και έχει έναν προπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια. Η Επιτροπή σας πάντοτε ε, μας υποστήριζε ε, όταν είχαμε κάποιο δημοσιονομικό αίτημα ε, στο παρελθόν και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και για να σας ενημερώσω, Πρόεδρε, και να ενημερώσω και τα μέλη της Επιτροπής, ε, στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, το 2010 θα είναι η τελική, το τελικό έτος όσον αφορά την αύξηση του προπολογισμού μας. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουμε ένα προπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ και ένα προσωπικό 350 ατόμων σε όλες τις κατηγορίες. Τα τελευταία 4,5 χρόνια ε, αρχίσαμε, είμαστε απόλυτα λειτουργικοί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας. Ε, έχουμε εφαρμόσει όλες τις ε, υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το καταστατικό του κέντρου και το τελευταίο και πέρυσι έγινε η πρώτη αξιολόγηση του κέντρου η οποία ολοκληρώθηκε και που αποδεικνύει ότι έχουμε μια σαφή παρουσία στο διεθνές ε, προσκήνιο. Τώρα θα με ρωτήσετε ποιος είναι ο ρόλος του ΕΚΠΕ, του Ευρωπαϊκού Αυτού Κέντρου. Ο ρόλος μας είναι, για να το πω απλά, είναι να προσφέρουμε στοιχεία και ενδείξεις σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να προσφέρουμε συμβουλές, πρακτικές συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη, να προσφέρουμε ε, κατάρτιση και πρακτική υποστήριξη στην, στα, στα ευρωπαϊκά όργανα και στα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να καταπολεμηθούν οι μολυσματικές ασθένειες. Τώρα, τα στοιχεία αυτά τα οποία προσφέρουμε εμφανίζονται με διαφορετικέ μορφέ. Όπω παραδείγματο χάρη εκθέσει επίβλεψη που αναλύουν τι τάσει σε διάφορες, διάφορων μορισματικών νοσημάτων. Ε, προσφέρουμε επιστημονικέ επιστημονικές ε, κατευθύνσει για τον έλεγχο ή την πρόληψη ε, εντοπίζουμε και διαδίδουμε τις καλές πρακτικές, ε, ε, εάν και εφόσον υπάρχει η διάδοση μιας νόσου, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, ε, αξιολογούμε τον κίνδυνο της απειλής, εάν και εφόσον υπάρχουν, έχουμε πολλά κρούσματα σε κάποια, για κάποιες νόσου, Όλη αυτή τη δουλειά ε, μπορείτε να την ε, δείτε και στο website μας, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Ένα άλλο πολύ, μια άλλη πολύ σημαντική δραστηριότητά μας ε, είναι η λειτουργία του, του, του, κέντρου πηγών των περιστατικών, αν θέλετε. Εδώ συλλέγονται πληροφορίες ε, από όλο τον κόσμο, 7 μέρες ε, την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο και προσπαθούμε να εντοπίσουμε ε, σημάδια για ε, αναδιόμενες απειλές της υγείας. Και αυτό το είδαμε και την, με την πανδημία της γρήπης όταν εμφανίστηκε τον Απρίλιο στην Βόρεια Αμερική. Μέσα από αυτό το κέντρο, το λειτουργικό κέντρο ε, συλλέξαμε τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία κοινοποιούμε στους συνεργάτες μας. Όμως δεν ασχολούμεθα μόνο με την ε, γρήπη αλλά και με 50 άλλες ε, ασθένειες γιατί δεν είναι και η μόνη απειλή δυστυχώς ε, την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επιστημονικά προγράμματα που καλύπτουν όλες αυτές τις ασθένειες, τις 50, τις 50 που ανέφερα και ε, συντονίζουμε και τη χρησιμοποίηση των, ε, ε, των εμβολίων, παραδείγματος χάρη για ασθένειες όπως είναι η φυματίωση, και οι πατήτηδες κτλ. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές μας προτεραιότητες, οι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας για φέτος. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν ε, στα, στις ασθένειε ασθένειες και την περαιτέρω ενδυνάμωση των συστημάτων για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Αναλύουμε τον, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αλλαγών του κλίματος στην διάρκεια διάδοση των μολυσματικών νοσημάτων στην Ευρώπη. Προσφέρουμε υψηλής επιότητας επιστημονικές συμβουλές και ε, κατευθύνσεις ε, σε, στα βασικά θέματα, στις βασικές ασθένειες που καλύπτει το ΕΚΠΕ και υποστηρίζουμε την ε, συλλογική απάντηση της Ευρώπης στην πανδημία της γρήπης. Ε, θα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση, Πρόεδρε, που αφορά την, τις αρμοδιότητές μας και τις ε, εντολές που έχουμε πάρει. Πρόεδρε, με την ε, άδεια σας θα ήθελα να προχωρήσω και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την πανδημία στην Ευρώπη, στην και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, ο νέος αυτός ιός είναι παρόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μια σταθερή ε, διάδοση σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα γεγονός άνευ προηγουμένου, τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν εξαφανίζεται η γρήπη. Ε, οπότε αυτό είναι μια προειδοποίηση ότι μπορούμε να περιμένουμε το φθινόπωρο. Εάν δείτε τα νούμερα και υποβάλλονται εκθέσεις ε, σε καθημερινό και αναφορές σε, καθημερινή βάση, επί του παρόντος έχουμε 46.000 ε, κρούσματα στην Ευρώπη επιβεβαιωμένα και 104 θανάτους. Όμως ε, στις χώρες ε, που έχουμε μεγάλο ρυθμό κρουσμάτων δεν γίνεται ο έλεγχος των νέων κρουσμάτων για το κατά πόσον είναι η νέα γρήπη ή όχι. Επομένως δεν έχουμε ασφαλή στοιχεία και δεν μπορούμε να, δώσουμε, να μιλήσουμε για αριθμούς. Οι χώρες που έχουν τα περισσότερα κρούσματα δεν μετράνε πλέον και αυτό συνέβη και στις ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη, στο παρελθόν. Επομένως, και και εμείς αλλά και οι Αμερικανοί έχουν πάψει να κάνουν ε, αναφορές και εκθέσεις, ε, να ε, κάνουν ανακοινώσεις καθημερινές, χρησιμοποιούν άλλα μέτρα. Τώρα, πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες πέρασαν από την πολιτική συγκράτηση στην πολιτική, ε, σε μια, πιο μετριοπαθή αν θέλετε πολιτική, ε, έτσι ώστε να περιορίσουν αν μη τι άλλο τον αριθμό των κρισμάτων. Να σας πω ότι μέχρι τώρα είχαμε 104 ε, επιβεβαιωμένους θανάτους, το οποίο είναι ένα ποσοστό όμως του των θανάτων, γιατί ε, όπως και για την εποχιακή γρήπη χρειαζόμαστε περαιτέρω ε, μελέτες για να έχουμε την σαφή και πραγματική εικόνα. Και συμφωνώ με την δόκτωρα Μάργαρετ Τσάν, που είναι η Γενική Διευθύντρια της, ε, του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι είναι μια μετριο, μέτρια πανδημία, μετριοπαθής πανδημία, όμως δεν είναι και τελείως αθώα. Τώρα, τι θα γίνει το φθινόπωρο στην Ευρώπη. Ε, φαντάζομαστε ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία που ακολουθήθηκε και στο νότιο ε, ημισφαίριο το καλοκαίρι, που γιατί εκείνη το χειμώνα για, την, για τους ε, για την Αυστραλία, την Αργεντινή, τη Χιλή. Επίσης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μελετήσαμε την κατάσταση στο νότιο ημισφαίριο πάρα πολύ προσεκτικά το φθινόπωρο και, το, και το χειμώνα, η γρήπη H1N1 θα είναι ο βασικός, ο κυρίαρχος ιός της, της γρήπης. Αλλά με θα διαμορφωθούν διαφορετικές εικόνες στις διάφορες χώρες. Γιατί οι κορυφές θα είναι διαφορετικές, αν θέλετε, ε, στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ε, οι, οι, αριθμοί ε, μέχρι στιγμής για την Ευρώπη είναι λίγοι. Δηλαδή εννοώ ότι έχει ε, ασθενήσει κάτω το 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Όμως το φθινόπωρο και το χειμώνα περιμένουμε ότι μέχρι το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, πληθυσμού συγγνώμη, θα μπορεί να μολυνθεί. Ε, αυτή όμως, ε, τονίζω, δεν είναι μια πρόβλεψη, απλώς είναι το χειρότερο σενάριο για την εξέλιξη του, του ιού. Και αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο, για το οποίο προετοιμαζόμαστε, ε, αν και εφόσον ο ιός και ο γενετικός, η γενετική ταυτότητα του ιού παραμείνει ως έχει και δεν μεταλλαχθεί και να γίνει πιο επιθετικός ή πιο βίαιος. Υπάρχουν όμως και πάρα πολύ καλά νέα. Καταρχάς η πρώτη καλή είδηση είναι ότι η ασθένεια αυτή είναι, δεν είναι πάρα πολύ σοβαρή, είναι ήπια, ε, όχι, δεν είναι τίποτα χειρότερο από μια κανονική γρήπη και αν δεν ε, αγχωθούν ε, οι άνθρωποι και δεν πάνε στην, στη δουλειά τους, δεν θα απουσιάσει και πολλοί κόσμος από, την, από τις δουλειές τους, άρα δεν θα διαταραχθούν οι βασικές υπηρεσίες. Επομένως, ε, για τις χώρες ε, που έχουν ένα πρόγραμμα συνεχούς παραγωγής ή συνεχούς εργασίας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τώρα, ποιο είναι τα, ποια είναι τα κακά νέα. Ότι η πανδημία αυτή θα ασκήσει μεγάλη πίεση στις υγειονομικές υπηρεσίες και στις, σε επίπεδο ε, παθολόγων, ας πούμε, αλλά και στις, ε, σε νοσηλευτικό επίπεδο. διότι Πάρα πολλοί ασθενεί, καταρχά θα θέλουν να δουν τον γιατρό του. Ε, και αυτός ο αριθμό ο των ασθενών που θα επισκέπτεται του ιατρού θα αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, ε, έστω και ένα μικρό ποσοστό αυτών που θα ασθενήσουν ε, χρειαστεί να νοσηλευτούν, αυτό σημαίνει ότι θα, θα υπάρχει μεγάλη πίεση και για τα νοσοκομεία, αλλά και κυρίω και για τι μονάδε εντατική θεραπείας. Επομένως, έτσι όπως και με τους προηγούμενους ε, ιούς πανδημίας, οι άνθρωποι που θα ασθενήσουν δεν θα είναι οι συνηθισμένοι ε, ασθενείς της κανονικής γρήπης, της εποχιακής γρήπης. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες δηλαδή ασθενών. Οι πιο ευάλωτοι είναι τα νέα παιδιά, οι ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι τα παιδιά μικρά παιδιά και οι έγκυες και αυτοί που έχουν κάποιες χρόνιες ασθένειες. Με την εποχιακή γρήπη ξέρετε ότι η ε, ηλικιωμένη τρίτη ηλικία, πάνω από τα 65 είναι αυτή που απειλείται περισσότερο. Τώρα, ποιες είναι οι εναλλακτικές ε, λύσεις που προσφέρονται. Και αυτό είναι επίσης μια καλή είδηση την οποία θα ήθελα να σας πω, είναι ότι είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την πανδημία σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές, με την Κομισιό, με την Επιτροπή σας εδώ και καιρό και είμαστε επομένως προετοιμασμένοι, καλά προετοιμασμένοι θα έλεγα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω ότι είμαστε η, καλύτερη, η καλύτερα προετοιμασμένη περιοχή του κόσμου ε, πολλές φορές μας ε, κατηγόρησαν ότι επενδύσαμε υπερβολικά για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, αλλά τώρα βλέπουμε ε, ότι απέδωσαν τα μέτρα αυτά. Τα περισσότερα κράτη έχουν, ένα, έχουν προγράμματα και είναι έτοιμα, έχουν, έχουν κάνει και κάποιες ασκήσεις, και έχουμε αναθεωρήσει ούτως ή άλλως, έχουμε εξετάσει συγγνώμη, όλα τα προγράμματα ετοιμότητας των κρατών μελών. Από το 2005 προετοιμαζόμαστε για, την, ε, για τις πανδημίες γενικότερα. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό σύστημα το οποίο λειτουργεί ε, και που αφορά την, τον συντονισμό και την κατανομή των, και την διάδοση των πληροφοριών. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα, επομένως, είναι να εξετάσουμε ε, αυτά τα σχέδια, η υπό το φως των γνώσεων που έχουμε για αυτό το νέο ιό και να δούμε αν χρειάζεται κάποια προσαρμογή ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, δεν θα πω ποια είναι όλα τα μέτρα τα οποία αφορούν αυτή την φάση, την ενδιάμεση φάση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ε, που μπορείτε να τις δείτε στο website μας. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και βιώσιμα. Υπάρχουν όμως ορισμένα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω, διότι αποτελούν προτεραιότητα για αυτούς που λαμβάνουν τι αποφάσεις. Το ένα είναι ότι θα πρέπει οι χώρες να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα υγειονομική περίθαλψης ε, έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό ασθενών και κυρίω τον, ε, τον βαριά ε, ασθενών που χρειάζονται εντατική Πρέπει να τετραπλασιαστεί ο αριθμό ας πούμε, κλινών στι εντατικέ ε, για να αντιμετωπίσουμε τα, τα, τα, τα, προβλήματα. Επίση, απλά μέτρα πρόληψη, όπω το να πλένουν τα χέρια του ε, και όσοι είναι άρρωστοι να μπαίνουν στο σπίτι του, ε, αυτά είναι απλά μέτρα τα οποία περιορίζουν τη διάδοση τη ασθένειας. Και αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια στο, στον κόσμο. Επίσης, από κάποια στιγμή, το φθινόπωρο ή το χειμώνα, θα έχουμε και το εμβόλιο και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας και πρόληψης. Βέβαια θα υπάρξουν πολλές ε, προκλήσεις με τα εμβόλια αυτά στην Ευρώπη. Ε, εμείς εξετάζουμε κάποια από αυτά τα οποία εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων μας. Τα εμβόλια για τη γρήπη είναι ασφαλή. Όμως, όταν χρησιμοποιηθούν, κυρίως ανάμεσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα υπάρχουν κάποιες παρενέργειες. Και συνεργαζόμαστε και με τον, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις Εθνικές Αρχές ε, για να ελέγξουμε τις, τις πραγματικές παρενέργειες που θα έχουν τα εμβόλια και για να μην ε, μας καταλάβουν εξαπίνεις ε, οι συνέπειες. Τώρα, να δούμε ποια είναι, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο. Καταρχά υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητε. Σα είπα κάποιες από αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλες. Παραδείγματο χάρη, ε, μήπως εμφανιστεί μια αντίσταση και μια αντοχή στα αντιϊκά φάρμακα. Ε, τι θα δώσει το μείγμα της εποχιακής γρήπης και της, του ιού της πανδημίας. Αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε τι θα γίνει. Στο νότιο ημισφαίριο το, τους χειμερινούς μήνες συμπεριφέρθηκε ο ιός αυτός πάρα πολύ καλά. Και το τρίτο είναι εάν αυτός ο ιός θα παραμείνει ήπιος αν θέλετε, όπως είναι τώρα. Και να μείνει σταθερός έτσι όπως είναι τώρα. Εάν δείτε το ιστορικό των προηγούμενων πανδημιών θα δείτε ότι ε, οι πανδημίες εξελίσσονται με πολύ ε, ε, διαφορετικό τρόπο. Και το, τα δεύτερο, το δεύτερο και το τρίτο κύμα είναι πιο παθογεν, παθογόνο, αν θέλετε, και πιο βίαιο από ότι το πρώτο. Πάντως αυτό το οποίο μας καθησυχάζει είναι ότι φαίνεται ότι ο τύπος αυτός ε, γρήπης, ε, αυτός ο ιός παραμένει σταθερός. Καθησυχαστικά σταθερός θα έλεγα. Και μέχρι στιγμής ε, δεν έχουμε, δεν έχουμε δει καμία αλλαγή στη σύνθεση του, του ιού. Αυτό είναι θετικό. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα να κάνουμε, Πρόεδρε, είναι να ολοκληρώσουμε την ετοιμότητά μας, λαμβάνοντα και τα ε, προγράμματα ετοιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη ε, μας όλες τις πληροφορίες ε, που έχουμε συλλέξει για τον ιό αυτό το τελευταίο, τις τελευταίες εβδομάδες και μετά χρειαζόμαστε αλληλεγγύη ανάμεσα στους πλώσιους, πλούσιους και στους λιγότερο, λιγότερο πλούσιους. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα εμφανιστεί και το φθινόπωρο, δηλαδή χρειάζεται μια αλληλεγγύη και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια. Αυτά Πρόεδρε, ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιάκοπ για αυτές τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσε. Ε, είμαι σίγουρος ε, πως θα υπάρξουν ε, πολλές ε, ερωτήσεις ε, από την πλευρά των συναδέλφων γιατί βέβαια το ζήτημα αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Να καλωσορίσω εδώ και επίσημα την Νέβα Μαγιόρη που είναι εκπρόσωπος της εκπροσωπεί το δικό μας και τον κύριο Ζακ Σέρες, τον πρόεδρο του της Επιτροπής Διαχείρισης του Management Board σας καλωσορίζω και σας θερμά. Και βέβαια, αν δεν υπάρξουν ε, πολλοί συνάδελφοι που θα θελήσουν να πάρουν τον λόγο, ε, θα μπορέσετε και εσείς να έχετε δυνατότητα να τοποθετηθείτε. Κυρία Γιάκοπ. Ε, προβήκατε σε μια ενημέρωση και σε μια παρουσίαση η οποία βέβαια δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Να δώσω λοιπόν καταρχήν τον λόγο στον συνάδελφο Πέτερ Λίζε που το ζήτησε και πρώτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Γιάκαμπ για αυτήν την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πρωτού ε, συζητήσουμε περαιτέρω και θέσουμε ερωτήματα, καταρχήν θα ήθελα να σας να συγχαρώ τον ε, κύριο Τζον Μπόουις, τον ε, πρώην συναδελφό μα ε, και συντονιστή από την πλευρά του ε, Κοινοβουλίου που είχε φροντίσει για τη δημιουργία ε, αυτού του κέντρου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πόλους και Ελέγχου Νόσων ε, και τώρα βλέπουμε πόσο απαραίτητο ήταν αυτό, αυτή η πρωτοβουλία που είχε ληφθεί. Τώρα, η ε, ισορροπία την οποία θα πρέπει να βρούμε εμείς τώρα είναι αυτή που θα πρέπει αφενός να λάβουμε υπόψη και να μην οδηγήσουμε βέβαια σε υπερβολικό πανικό α, τους πολίτες με στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν ακόμα ε, υποστηριχθεί με τα κατάλληλα δεδομένα και αφετέρου βέβαια να μην υποτιμήσουμε υπερβολικά την κατάσταση. Είναι μια ισορροπία λοιπόν την οποία θα πρέπει να επιτυχάνουμε κάθε μέρα εκ νέου. Ε, ειδικότερα οι χώρες με ε, ιδιαίτερα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας παρατηρείται μεγάλη εξάπλωση, αλλά και σε άλλες χώρες συμβαίνει το ίδιο. Για παράδειγμα στη Βραζιλία έχουμε εκατοντάδες νεκρούς Πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι ε, οι περισσότερες ασθενείς κατά τις 78 πρώτες ώρες ε, που νοσούν και στις οποίε είναι κέρια η παρέμβαση ιατρική δεν ε, πηγαίνουν σε γιατρό. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό, δηλαδή η ιατρική ε, Όμως θα ε, θα συμφωνήσω με τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος του CPM, e, δηλαδή ε, ο κ. Μοντγκόμερ, ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης. Ε, εμείς έχουμε ε, φτάσει στο σημείο από την πλευρά της Γερμανίας που είχαμε πει ότι για το 50% μπορούν τα ταμεία της δημόσιας υγείας να ε, ε, χρηματοδοτήσουν τα εμβόλια, αλλά όχι για το υπόλοιπο 50% και θα πρέπει να δούμε τις άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αλλά βέβαια ε, δεν υπάρχει ρεαλιστικό ενδεχόμενο να έχουμε μόλυνση πάνω από 50% του πληθυσμού. Όμως ε, θα ήθελα να αναφέρω επανειλημμένα ε, το γεγονός ότι το, οποίο έχει μάλλον παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι νοσούν εύκολα τα παιδιά και η κυρία Γκρουστέ το έχει αναφέρει και αυτό επανειλημμένα. Δηλαδή οι συστάσεις ε, συχνά οι οποίες γίνονται για τους ενήλικες δεν ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για τα παιδιά. Και αυτό για παράδειγμα και σε σχέση με τα φάρμακα. δεν έχουμε για παράδειγμα ένα αντιϊκό φάρμακο αυτή τη στιγμή το οποίο να διατίθεται και με τη μορφή χυμού. Ε, δηλαδή, αν ε, ζητήσουμε από τους γονείς να δημιουργήσουν ε, ένα σκεύασμα μόνοι τους χρησιμοποιώντας το φάρμακο σε άλλη μορφή, πολλές φορές δεν το κάνουν, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν σωστά. Άρα λοιπόν, πέραν από αυτό, υπάρχει και το ζήτημα του κατά πόσο έχουμε να κάνουμε μια υποψία, δηλαδή με μια εκτιμόμενη περίπτωση. Ε, και του πώς χαρακτηρίζουμε μια τέτοια. Δηλαδή, ε, ε, εάν πούμε ότι οποιοδήποτε άτομο έχει πυρετό, εκδηλώνει πυρετό πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου θα πρέπει να έχουμε μετά προστατευτική ένδυση και ούτω καθεξής, καλώς. Αλλά για παιδιά κάτι, δεν μπορεί, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με αντίστοιχο τρόπο. το ίδιο ισχύει και για τον εμβολιασμό. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί ε, ούτως ώστε να μην προβούμε σε υπερβολικές συστάσεις. Υπήρξε μια σύσταση από την πλευρά της Υπουργού Υγείας, η οποία εκ των υστέρων μας είπε ότι ήταν προσωπική άποψη, σύμφωνα με την οποία ε, με βάση κάποιες μελέτες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα θα πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά όχι τώρα αλλά την άνοιξη. Εγώ δεν μπορούσα να βρω κανέναν άλλο εμπειρογνώμονα ο οποίο να μου πει το ίδιο, ότι θα πρέπει δηλαδή τα παιδιά να εμβολιαστούν την άνοιξη. Ε, Εσεί ίδια το είπατε μόλι τώρα, ότι αν υπάρξει πρόβλημα θα υπάρξει το φθινόπωρο ή το χειμώνα, όχι την άνοιξη. Άρα λοιπόν παιδιά, ειδικότερα στις ομάδες κινδύνου θα πρέπει να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατό. Και θα θέλαμε κι εσείς να επιστήσετε την προσοχή σε αυτά τα ζητήματα για μία ακόμα φορά. Επίση, σε ό,τι αφορά ε, τι κλιματικέ μεταβολέ και τι μολυματικέ ασθένειε, μα είπατε ότι θέλετε να κάνετε κάτι σε σχέση με το δικό σα ε, ε, πρόγραμμα εργασία. Ε, θα θέλαμε όμω να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Προλέπετε να κάνετε κάτι, γιατί βέβαια αυτό το ζήτημα θα μα ασχολήσει πάρα πολύ μέσα στου ερχόμενου μήνε στη δική μα επιτροπή. Αν έχετε λοιπόν κάτι από τη δική σα πλευρά που προβλέπετε να κάνετε, θα θέλαμε να το ακούσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Πέτερ Λίζε. Η ακόμα Ροτ Μπέρεντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω γεια σου Φρανκ στον συνεργάτη μου από το Ελσίνκι. τώρα, Κυρία Γιάκα, ε, σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας ε, παρουσιάσατε σήμερα εδώ. Έχω κάποια ερωτήματα να θέσω. Ε, κάποια πραγματικά από τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι με άφησαν κατάπληκτη. Ε, καταρχήν, προφανώς έχουμε να κάνουμε μια επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια, αλλά δεν είναι η πρώτη επικίνδυνη λεωδική ασθένεια και η πρώτη επικίνδυνη γρήπη την οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε μέσα στα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν σε κάποια κράτη-μέλη διαπίστωσα το εξής. Αφενός σε πάρα πολύ ε, υψηλό βαθμό πανικού και ταυτόχρονα ε, μια κατάσταση σοκ, δηλαδή πλήρους απραγίας. Θα ήθελα να ακούσω από τη δική σας πλευρά τι γίνεται. Σε μια περίπτωση όπου πραγματικά υπάρχει φόβος ε, πανδημίας για την ε, λήψη απλών μέτρων υγιεινής. Απλών μέτρων υγιεινής. Γιατί δηλαδή πρέπει θα πρέπει 20 ε, άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ένα κουμπί σε ένα σανσέρ ή χρησιμοποιούν ένα χερούλι μιας πόρτας να είναι σε θέση να διαδώσουν τον ιό σε χιλιάδες άλλους. για παράδειγμα, σε συνδρομικού σταθμού, σε αεροδρόμια, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε κοινοβούλια, σε δημόσιου χώρου, ε, να, να υπάρχουν παντού δυνατότητε απολύμανση των χεριών. Κάποια ενημέρωση, ούτως ώστε δηλαδή να έχουμε κάποια απλά μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται και ούτω ώστε να κάνουμε κάτι σε ένα πρώτο επίπεδο για να αποφύγουμε να προλάβουμε την περαιτέρω διάδοση τη ε, ασθένεια. Ε, υπάρχουν και άλλε δυνατότητε. Ο κύριο Λίζε το ανέφερε μόλι τώρα. Γιατί δεν υπόθηκε με σαφήνεια ποια είναι τα συμπτώματα. Γιατί, η πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύθηκε περισσότερο. Δηλαδή, πότε θα πρέπει να θεωρούμε κάποιον ύποπτο ότι έχει νοσήσει συμπτώματα. Συγκεκριμένα, πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου ε, για ενήλικες, αλλά όχι σίγουρα για τα παιδιά, γιατί ε, ε, τα παιδιά μπορούν να νοσήσουν επανειλημμένα μέσα σε ένα χρόνο με πυρετό πάνω από 38 βαθμούς και δεν μπορούμε κάθε φορά να τα θεωρούμε ως ύποπτους, ως ύποπτες Δηλαδή, γιατί δεν υπήρξε μια καλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή, η έλλειψη πρόληψης, η έλλειψη precaution. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν μας βοήθησε αυτό. Και μάλιστα, σε ορισμένε περιπτώσεις, ε, δημιουργήθηκε πανικός και τίποτα άλλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, ε, τα εμβόλια, πέρα από την ε, των χείρων έχουμε βέβαια και την κανονική εποχική γρήπη η οποία θα μας βρει. Α, δηλαδή θα έχουμε δύο διαφορετικά είδη γρήπης τα οποία είναι ιδιαίτερα μολυσματικά και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα για τις ευπαθείς ομάδες. Τι προτείνετε εσείς για αυτές τις ευπαθείς ομάδες, γιατί οι συστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικές. Κάποιοι λένε δηλαδή ότι αυτά τα άτομα θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά της γρήπη αυτής. Κάποιοι άλλοι λένε όχι να εμβολιαστούν μόνο κατά της κανονική εποχιακή γρήπη. Τι τελικά πρέπει να κάνουν. Επίσης, ε, θεωρούμε προφανώς ότι τα εμβόλια αυτά είναι ασφαλή, αλλά ε, ειδικότερα τα νέα εμβόλια τα οποία έχουν, ε, έχουν κατασκευαστεί, ε, έχουν παρασκευαστεί ε, τόσο γρήγορα, δεν ήταν δυνατόν να συνοδευτούν και από κατάλληλε ε, κλινικές μελέτες. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη, ήδη σε ό,τι αφορά τη διάθεση των αντιοικών, δεν λειτουργεί εδώ και άρα δεν λειτουργεί και σε σχέση με ένα τέτοιο ζήτημα η Επιτροπή έχει τα ε, απαραίτητα κονδύλια στη διάθεσή της, ε, εκείνη τα διαθέτει, οπότε το μόνο που μπορούμε να βασιστούμε εδώ είναι η λογική των άλλων κρατών μελών. Ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας, που είσαστε εδώ μαζί μας ε, σήμερα το απόγευμα. Να σας κάνω μια διπλή ερώτηση, αν θέλετε. Το ένα αφορά την μέθοδο εργασίας ε, της υπηρεσίας σας, του οργανισμού σας. Πώς ε, επιλέγετε τους εμπειρογνώμονές σας, ποιο είναι το καθεστώς τους, ποιος, ποιες, είναι, ποιες είναι οι μέθοδοι εργασίας και συνεργασίας μαζί τους και συμμετέχετε στις εργασίες ε, με ποιο τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την επιτροπολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσει από τι πολιτικέ αρχέ. Αυτό ήταν το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά πιο συγκεκριμένα την γρήπη και το εμβόλιο. Καταλάβαμε ε, ότι αντιμετωπίζουμε, είμαστε ανάμεσα στη σκύλα και στη Χάριβη, αν θέλετε. Το ένα είναι εάν και εφόσον εμβολιάσουμε να γίνει μέσα στις προθεσμίες από τη μια και από την άλλη ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τις ε, άμεσες ή έμεσες συνέπειες της παρενέργειας των εμβολίων. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς ε, την επίλυση αυτών των δυσκολιών που δεν είναι και λίγες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είναι εδώ η κυρία Και εγώ έχω πολλές ερωτήσεις να υποβάλω. Μας παρουσιάστηκε αυτή η πανδημία, ενώ οι αριθμοί, όπως αναφέρατε και εσείς, 46.000 περιπτώσεις, 104 θάνατοι. 104 θάνατοι είναι πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας χωρίς να έχουμε και εμβόλιο. Δεύτερον, όταν γίνεται εμβολιασμός, πάντα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το όφελος και η βλάβη καμιά φορά. Ποια είναι τα ωφέλη από, μια τέτοι, από ένα τέτοιο είδους εμβολιασμό μιας ε, μέτριας εμβέλειας πανδημίας. Ή δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός αυτό ο ιός, ή είναι πολύ μεταδοτικός. Τώρα, όσον αφορά τους κινδύνους, το ρίσκο. Εγώ είχα πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά της ε, υπατήτηδας Β. Σκέφτομαι τον νόμο Κουσνέρ στη Γαλλία που ζητάει να υπάρχει σαφέστατη και ελεύθερη ενημέρωση. Δεν έχουμε τέτοιου ενημέρωση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε ποια είναι τα συστατικά του εμβολίου. Εάν πρόκειται για προσθετές ουσίες που περιέχουν αλουμίνιο, ξέρετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ε, εάν έχουμε άλλες ουσίες ε, στις οποίες περιέχεται υδράριος, επίσης υπάρχει κίνδυνος. Στη φορμαλδεΐδη επίσης υπάρχουν άτομα τα οποία είναι αλλεργικά. Και άλλες ουσίες τέτοιες επικίνδυνες μπορεί να περιέχονται. Το ερώτημα μου είναι, έχουμε αρκετή εμπειρία επί του θέματος και χαίρομαι που είστε εδώ, για να μπορέσετε να μας πείτε ότι ελτερεύουσες επιπτώσεις που θα έχει για την υγεία κάποιο εμβολιασμό είναι τόσο μικρές σε σχέση με το όφελε. Επίσης, ανάλογα με τα, αν πρόκειται για την Σανοφή, την οβαρτή, έχουμε διαφορετικά συστατικά. Όπω το ασπράδι αυγού. Έχουμε άτομα τα οποία είναι αλλεργικά στο ασπράδι, αλλά τα οποία είναι σε κάποια αλλεργικά σε ζωικά κύτταρα. Πείτε μας λοιπόν εσείς τι συμβαίνει. Εμεί πρέπει να σας πω ότι στη Γαλλία παραγγείλαμε κάποια εκατομμύρια δόσεις. Θα γίνει λοιπόν μαζικός εμβολιασμός στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Το ερώτημα είναι, έχουμε αρκετή εμπειρία για τις ε, κρίσιμες πληθυσμιακές ομάδες, για τις ευαίσθητες. Διότι εδώ λέει ότι όλοι οι ιατρικοί κύκλοι λέγουν να εμβολιαστούν οι πάντες. Μία νοσοκόμα που είναι έγκυος, μία ιατρός που είναι έγκυος. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι εάν εμβολιαστεί δεν θα επηρεάσει το έμβριο. Δεν θα επηρεάσει το έμβριο. Ξέρουμε αν ο εμβολιασμός σε σχέση με τον υδράργυρο, το αλουμίνιο, δεν θα επηρεάσει το έμβριμο. Έχουμε αρκετή πείρα. Ξέρουμε ποιε θα είναι οι άλλε επιπτώσει και μα λένε όλοι γρήγορα, γρήγορα, να πάτε γρήγορα. Αυτό το ακούμε παντού. Ποια είναι τα ωφέλη. Αυτή τη στιγμή πολλά άτομα ε, έχουν ε, γρήπη και ε, έγιναν καλά. Και οι παίκτε του Ράγκμπι στη Γαλλία και άλλοι. Μετά, ποιος θα είναι υπεύθυνο. Και εδώ η ερώτηση πάει στην Ευρώπη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα δώσει το πράσινο φως για να τεθεί το εμβόλιο στην αγορά. Από νομικής πλευράς μέχρι σήμερα ξέραμε ότι αυτή η εξουσιοδότηση διάθεση στην αγορά διδόταν από κάθε χώρα χωριστά. Οι διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες ξέρουμε ότι ζήτησαν στη ΣΥΠΑ να ε, αποποιηθούν τις ευθύνες των ε, δυσκολιών που θα προκύψουν ενδεχομένω ή των προβλημάτων θα προκύψουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εμείς όπως ξέρετε είπαμε στη Γαλλία έχουμε παραγγείλει σχεδόν μία, ένα εμβόλιο για κάθε Γάλλο. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις χορήγηση αυτού του εμβολίου. Το 1976 στη είπα πρέπει να σας πω ότι ε, πέθανε ένα στρατιώτης από αυτή την γρήπη εμβολιάστηκε το 40% του πληθυσμού με πρόεδρο το Φόρτ εξαιτίας των ε, αρνητικών επιπτώσεων ε, μετά από τρει μήνε σταμάτησε ο εμβολιασμό και διερωτώμε. Μήπως μήπω βιαζόμαστε, μήπω ζητούμε να γίνει μαζικό εμβολιασμό χωρί να έχουμε εξετάσει ποιε θα είναι οι δευτερεύουσε και αρνητικέ επιπτώσει. Σα ευχαριστώ. Έχει τεθεί επανειλημμένα αυτό το ερώτημα από του συναδέλφου θα έχετε δυνατόν να απαντήσετε. Έχουμε την κυρία Μαριάννα Γιανακουδάκη τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Γιάκαμπα για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ε, και θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της, ε, του εμβολιασμού για την εποχιακή γρήπη. Παρά τους, ε, την στόχο του να επιτευχθεί το 75% σε επίπεδο εμβολιασμού σε ό,τι αφορά έως το 2010. Οι περισσότερες χώρες έχουν μείνει πολύ κάτω από αυτό το όριο. Η Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε μια πρόταση για συστάσεις του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την εποχιακή γρήπη με στόχο την ε, αύξηση της κάλυψης του εμβολιασμού μέχρι αυτόν τον στόχο και να ε, θέσει μια αντίστοιχη αξίωση για τα εθνικά σχέδια δράσης. Όμως αυτή η πρόταση ε, δεν ε, καλύπτει και την ανάγκη για την καλύτερη ενημέρωση και την κοινή χρήση των πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και των κρατών μελών. Οπότε σας ρωτώ, θα μπορούσε το ECDC να αναλάβει εδώ ένα πιο ενεργητικό ρόλο όπως το έπραξε και σε σχέση με τον εμβολιασμό για τη γρήπη H1N1 προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά ε, την εποχιακή γρήπη και μπορούμε να βασιστούμε στα στοιχεία τα οποία ε, έχουν συλλεχθεί από τις διάφορες ε, περιοχές και τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τους δικούς τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και εγώ έχω με τη σειρά μου να θέσω ένα-δύο ερωτήματα. Είπατε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν εκπονήσει δικά τους σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης. Έχουν ε, όλα την ίδια ποιότητα αυτά τα σχέδια δράσης. Υπάρχει ένα ελάχιστο αν θέλετε ένα ελάχιστο κοινό ε, παρονομαστή, ή απλά ε, έχετε κάποια γενικά σχέδια και μετά δεν ξέρετε τι ακριβώς θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, Επίση, θα ήθελα να ακούσω πόσες εταιρείε, πόσες φαρμακομηχανίες παράγουν αυτό το εμβόλιο. Εγώ ακούω πάντα για δύο, ε, οι οποίε νομίζω είναι γερμανικέ. Μήπω ε, υπάρχουν παραπάνω. Αν λέτε ότι έω και ένα τρίτο του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσβληθεί, μιλάμε για 150 εκατομμύρια άτομα και αν θα πρέπει να γίνει δύο φορέ ο εμβολιασμό για αυτά τα άτομα, μιλάμε για 300 εκατομμύρια δόσει εμβολίου ε, θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο και πόσο γρήγορα θα μπορούσε να παραχθεί ένα τέτοιο αριθμό εμβολίων. Ε, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα τα εμβόλια. Θα έρθουν σε ένα, ενδεχομένως σε, μια, σε ένα δεύτερο, σε ένα, τρίτο στάδιο η φάση παραγωγής. Ο λόγος σε, σε εσάς ε, για να απαντήσετε κύριε Διάκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής για την ε, υποστήριξή σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα που μου θέσατε. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν να συνοψίσω ε, τις απαντήσεις που θα σας δώσω. Θα ήθελα καταρχήν να ε, επενθυμίσω πως ο Τζον ε, στην προηγούμενη Επιτροπή Περιβάλλοντος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να υποστηρίξει τις αρχικές δραστηριότητες του ECDC και σας ευχαριστούμε πολύ που υπενθυμίσατε τη πολύ σημαντική δουλειά που έκανε για να υποστηρίξει το ECDC και ε, όπως είπα και στην παρουσίαση μου Ελπίζω πως και εσείς ε, θα ορίσετε ένα ε, σημείο επαφή, έναν αρμόδιο για την επαφή με το ECDC, κάποιον ο οποίος θα είναι αρκετά ε, εδώ γνωστός ώστε να μπορεί να βρίσκεται σε επαφή με όλους σας και να έρχεται συνεχώς σε επαφή μαζί μας. θα ήταν πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπερβολική αντίδραση ή τον πανικό ο οποίος προκλήθηκε σε κάποια κρατημέλη και το οποίο ε, θέσατε. Ε, ε, είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν είχα την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε τόσο πανικός όπως τότε με το 2005 και την γρήπη των πτηνών. Όταν δηλαδή βλέπαμε πως προσέγγιζε τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πραγματικά υπήρξε ε, πανικό. Ε, είχαμε δει δηλαδή την εποχιακή γρήπη, την γρήπη των πτηνών και την ε, γρήπη των χείρων που είδαμε ότι πράγματι τελικά μπήκε εντός των συνόρων της Ευρώπης Αλλά ε, πράγματι ήταν καλό το ότι υπήρξε όλη αυτή η συζήτηση και στο δημόσιο επίπεδο ε, για τη γρήπη γενικά. Οπότε τώρα που τελικά βρέθηκε εδώ, εντός δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεν υπήρξε τόσο εκτεταμένος ε, πανικός. Αλλά πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η συζήτηση με το ευρύ κοινό σε ό,τι αφορά τη γρήπη. Υπάρχουν όλες οι γνώσεις σε ό,τι αφορά τα όσα θα πρέπει να κάνει ο πολίτης. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα πλήση υγιεινής που θα πρέπει πρέπει να λαμβάνουν όλοι ή για παράδειγμα τα, τα τα ζητήματα κοινωνική πρόληψη, δηλαδή ότι όποιο ασθενεί θα πρέπει να μένει στο σπίτι του ή να στέλνεται στο σπίτι του από το χώρο εργασία του. Ε, ε, θέλουμε να συνεργαστούμε εδώ στενά με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και ένα δίκτυο ενημέρωση το οποίο ε, ναι, μεν. Ε, ε, λειτουργεί υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ε, και στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να διαφανίσουμε ότι και τα κράτη-μέλη θα θέσουν ενεργά αυτό το ζήτημα στη δική τους ε, ατζέντα και την ενημέρωσή του ευρέως Και ο ρόλος του ECDC κατά την άποψή μου εδώ είναι ακριβώς να να κρατά συνεχώς ενήμερα τα τα κράτη-μέλη ε, και, το, ε, και την ε, Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις ενημερωμένες νέες πληροφορίες και πάντα να παρέχει υποστηρικτικό, υποστήριξη. Τώρα, πολλοί από εσά θέσατε ζητήματα σε σχέση με τον εμβολιασμό και αντιλαμβάνομαι πλήρω το γιατί τα θέσατε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω λοιπόν συνοψίζοντας σε ένα δεύτερο ζήτημα της απαντήσης που θα δώσω. Καταρχήν έχουμε τα δύο συμβόλαια μεταξύ, ε, δηλαδή αυτό της εποχιακής γρήπης και αυτό της, ε, ε, του H1N1. Εμείς υποστηρίζουμε το να εστιάσουμε στον εμβολιασμό για την εποχιακή γρήπη και μόλις είναι διαθέσιμο το εμβόλιο για την νέα γρήπη, το οποίο αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να είναι διαθέσιμο, να ακολουθήσετε τη δική σας στρατηγική σε ό,τι αφορά την εποχιακή, τον εμβολιασμό και την εποχιακή γρήπη. Για να καλύψετε τις δικές σας δηλαδή ευπαθείς ομάδες. Μιλάμε δηλαδή για ε, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, για άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα άνω των 65 ετών. Αυτές είναι ευπαθείς ομάδες και για αυτές θα πρέπει να προχωρήσετε με τον εμβολιασμό για την ε, ε, εποχιακή γρήπη. Άλλωστε, τον λόγο εμβόλιο είναι απολύτω ασφαλέ. Πάντα για την εποχιακή γρήπη. Ε, αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι έχει θέσει ένα στόχο η 85% ε, νομίζω πως είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει 75% ε, κάλυψη σε ό,τι αφορά τους, ε, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με χρόνες παθήσεις και να σας πω ότι κάναμε μία μελέτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς έχει η κατάσταση και διαπιστώσαμε ότι στις 27 χώρες, σε 27 κράτη-μέλη, μόνο δύο επιτυγχάνουν αυτό το στόχο, καλύπτουν δηλαδή αυτό το στόχο και άλλα τρία κράτη-μέλη είναι σχεδόν ε, πληρούν αυτό το στόχο και μόνο 10 κράτη-μέλη ε, μας διαβιβάζουν και μας ε, δεδομένα σε ό,τι αφορά την κάλυψη του εμβολιασμού σε ό,τι αφορά την εποχιακή γρήπη. Άρα λοιπόν είναι καλό το γεγονός ότι προέβη σε αυτήν την κοινοποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να τεθεί αυτός ο στόχος δηλαδή της αύξησης της κάλυψης εμβόλια Και προφανώ ε, εμεί ε, θα με τα χαρά θα αναλάβουμε ένα συντονιστικό ρόλο εδώ, όπω έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να γίνει αυτό ο διαγωνισμό μεταξύ εμβολίου κατά εποχιακή γρήπη και κατά H1N1. Ε, το εν λόγω εμβόλιο για το H1N1 δεν είναι ακόμα διαθέσιμο. Και αυτό το εμβόλιο για του υγιεί ενήλικε, επαναλαμβάνω υγιεί ενήλικε, βρίσκεται ακόμα σε φάση κλινική δοκιμή, η οποία θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές ή μέσα Οκτωβρίου. Τότε η Ειδική Επιτροπή της, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα θα έχει αναλάβει τις εργασίες της και θα μπορέσει να λάβει ε, μία απόφαση ως προς το κατά πόσο θα διοδοτήσει το λόγο εμβόλιο ή όχι και εκεί βέβαια θα ληφθούν υπόψη και όλες οι παρενέργειες οι οποίες θα έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της, των κλινικών δοκιμών. Άρα λοιπόν αναμένουμε την αδειοδότηση ε, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, τότε θα αρχίσει λοιπόν να βγαίνει πλέον ε, στη διάθεση ε, το εμβόλιο τύπου, για τον τύπο H1N1, αλλά μόνο για τους υγιείς ενήλικες, για τις τρεις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή για τα παιδιά, για τις εγγύους και για άτομα με χρόνους παθήσεις, θα έχουμε στη συνέχεια την έναρξη ε, των κλινικών δοκιμών. Άρα λοιπόν για παιδιά δεν υπάρχουν ακόμα τέτοιου είδους κλινικές δοκιμές και άρα λοιπόν για τις ιδιαίτερα φαθείς ομάδες, για τα risk groups θα αργήσει περισσότερο το εμβόλιο. Ε, και μπορεί να έρθει το εμβόλιο μόνο αφού θα έχουν ολοκληρωθεί αντίστοιχε κλινικές δοκιμές. Ε, κάποιοι με ρωτήσατε ε, επιχειρήσεις υπάρχουν εσείς ε, Πρόεδρε, ναι. Έχουμε κάποιες ε, πολυεθνικές αλλά και κάποιες εθνικές επιχειρήσεις οι οποίες ε, παράγουν εμβόλια για τη δική τους χώρα αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις βέβαια ισχύει η εθνική νομοθεσία που καλύπτει τις φαρμακοβιομηχανίες και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάλυψη από την EMEA σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτές τις εθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Τώρα, ακόμα ε, και αν ε, ε, όταν θα διοδοτηθεί και θα, το εμβόλιο και θα παράγεται σε μαζική κλίμακα, προφανώς θα υπάρξουν παρενέργειες. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά με τα εμβόλια γρήπης. αλλά ε, εν γέννη τα εμβόλια γρήπης ε, έχουν παρουσιακά ε, αποδειχθεί ασφαλή, δεν έχουμε δει πολλές επανενέργειες και η δική μας αρμοδιότητα του ECDC είναι να παρακολουθούμε ακριβώς την κατάσταση. Όταν θα ξεκινήσει λοιπόν η μαζική χρήση των εμβολίων, ο μαζικός εμβολιασμός, θα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης ώστε να παρακολουθούμε την κατάσταση για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε παρενέργειες προκύψουν. Αυτά λοιπόν ως απάντηση σε σχέση με τα όσα ερωτήθηκαν σε σχέση με το ζήτημα του εμβολιασμού. Τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια άλλα ζητήματα. Πέτρε ε, ε, μου ζήτησατε να αναφερθώ στην ε, σχετική στρατηγική ε, απομόνωση στη Γερμανία. Άρα λοιπόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό προσπαθεί να κάνει η Γερμανία είναι να μειώσει την εξάπλωση του ιού απομονώνοντας ε, τις ε, νέες εμφανιζόμενες ε, περιπτώσεις, τα νέα κρούσματα. Ε, όλες οι χώρες βρίσκονται αρχικά σε αυτή τη φάση, αλλά όπως ε, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων, ε, περνούν στο, στην επόμενη φάση οι χώρες δηλαδή από την, ε, από την, ε, από την απομόνωση περνάνε πλέον στην, ε, στην μείωση του αντικτύπου στην, της πανδημίας που, συνοδεύει, που συνοδεύεται συγγνώμη, από διαφορετικών, διαφορετικού είδους μέτρα, όχι δηλαδή με μέτρα όπως η απομόνωση. Η Γερμανία βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη φάση της απομόνωσης και μια πιθανή εξήγηση είναι ότι προσπαθούν ε, να προλάβουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού ε, για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι ακόμα διαθέσιμο το εμβόλιο. Περιμένει δηλαδή κανείς μέχρι να είναι διαθέσιμο το εμβόλιο και στη συνέχεια ξεκινάει μαζικά τον εμβολιασμό. Και μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτά τα δύο στάδια προχωράει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή περνάει πλέον στο mitigation, δηλαδή στη μείωση του, των συνεπειών από, ε, από την εξάπλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα, σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη δημοσιότητα ε, για τα μέτρα, πρακτικά μέτρα υγιεινής ε, που ανέφερε η κυρία Ντάκμα Μπέρεν σε άλλη επιτροπή είχα ε, αναφέρει αυτό το παράπονό μου ότι δεν έχουμε αυτά τα αντισηπτικά προϊόντα όταν ε, ε, ταξιδεύω στην Ασία, δεν βλέπω μόνο αυτές τις μάσκες, έχουμε παντού αυτά τα αντισηπτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για, για τα χέρια του. Ε, νομίζω πως ε, μπορούμε να εργαστούμε σε σχέση με αυτό, να συνεργαστούμε και ε, να, το, να γίνουν κάποιες συστάσεις στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή. Υπάρχει βέβαια εδώ κάποιο κόστος, αλλά η καλύτερη πρόληψη είναι πραγματικά αυτό, δηλαδή να πλένει κανείς τακτικά τα χέρια του και να μην αγγίζει το πρόσωπό του, το στόμα του με τα χέρια του, γιατί αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να εισέλθει ο ιός μέσα στο σώμα. Ε, συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εργαστούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι μάσκες, δεν έχουμε βρει ακόμα επιστημονικέ ενδείξει επιστημονικά στοιχεία για το ότι είναι αποτελεσματικέ. Δεν είμαστε ιδιαίτερα κατά, αλλά ούτε είμαστε ε, υπέρ. Ε, κάποιες ε, χώρε είναι υπέρ της χρήσης τη μάσκα, αλλά εμεί εξετάσαμε τα επιστημονικά στοιχεία και δεν δικαιολογείται, δεν υπάρχει κάτι που να τεκμηριώνει πράγματι την, τη χρήση της μάσκας, αλλά εάν κάποια θεωρήσουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες, δεν έχουμε κάτι εναντίον τους. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ε, ενημέρωση. Επίσης η Ντάκμα Ροντμπέρεντ με ρώτησε ως προς το ποιες συστάσεις θα έδινα σε ό,τι αφορά την εποχιακή γρήπη. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι ότι μόλις διατεθεί στην αγορά ε, το ε, εμβόλιο για την εποχιακή γρήπη, παρακαλώ πηγαίνετε, εμβολιαστείτε και όταν θα διατεθεί το ε, εμβόλιο για το H1N1 θα εξαρτηθεί από την δική σας εθνική στρατηγική. Η δική μας ε, σύσταση είναι να ξεκινήσει άμεσα μόλις θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο για τις ομάδες ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Βέβαια για αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου είπαμε ότι θα είναι λίγο αργότερα διαθέσιμο το εμβόλιο. Αλλά καθώς η ε, τα, οι σχετικέ στρατηγικέ βρίσκονται πλήρω στα χέρια των 100 μελών, αποτελούνται δηλαδή εθνική και όχι κοινοτική αρμοδιότητα, μπορούν τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν κατά πόσο θα επεκτείνουν τον εμβολιασμό στο σύνολο του πληθυσμού ή, αν θα περιορίσουν τον εμβολιασμό ε, στι ε, ομάδε υψηλού κινδύνου. συνήθω οι χώρε εκείνε οι οποίε έχουν τα κονδύλια για να ε, προβούν σε αυτόν τον εμβολιασμό μπορούν συνήθω το κάνουν και υπάρχει και αυτή ε, βέβαια υπάρχει ε, το, το, επιχείρημα ε, υπέρ του εμβολιασμού ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει μια μετάλλαξη του ιού σε ένα πιο μολυσματικό τύπο. Και επίσης θεωρούμε πως ένας, ένα μικρό μέρος αυτής της της ανοσίας που υπάρχει ήδη στον πληθυσμό οφείλεται ακριβώς σε ένα, σε ένα ε, μαζικό εμβολιασμό που είχε γίνει κατά τα ε, δεκαετία του 1950. Οπότε Ε, θα μπορούσε ένα τέτοιο μαζικότερο εμβολιασμό να σα βοηθήσει να καταπολεμήσετε ακόμα καλύτερα την εξάπλωση του ιού. Σε ό,τι αφορά τι ε, μεθόδου εργασία, ε, σα ευχαριστώ πολύ για τη σχετική ερώτηση, δηλαδή του πώ επιλέγουμε του εμπειρογνώμονέ μα. Εδώ ακολουθούμε πάντα την ε, προσέγγιση, την πολιτική της διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούμε και τα όσα βλέπει το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, διορισμό όχι μόνο του προσωπικού μας αλλά και τους, ε, των εμπειρογνωμών μας. Όλα, λοιπόν, όλοι, όλες τις δημοσιεύονται εκεί. Ε, και γίνεται κανονικά διαδικασία. Τώρα, το καθεστώ ε, μπορεί να είναι διαφορετικό για αυτού του επιστήμονε, δηλαδή μπορούν να είναι ε, μόνιμα, τακτικά δηλαδή μέλη επιστημονικών επιτροπών ή μπορεί να εργάζονται για μα ανεξάρτητα ω εμπειρογνώμονε, αλλά σε κάθε περίπτωση για μα είναι απαραίτητο ε, να έχουμε μια διαφανή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους ε, συμβούλους. Ακολουθούμε και πάλι το καταστατικό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους ειδικού επιμονόμενου, το χρησιμοποιούμε μόνο όταν υπάρχει μια ομάδα εργασίας η οποία έχει συσταθεί μετά από το λίτο του Διοικητικού μα Συμβουλίου και για το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, να, έχουμε και έναν, δύο ειδικού εμπειρογνώμονε η αμοιβή για αυτού ε, πάντα αποφασίζεται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Ποτέ, δηλαδή, ποτέ δεν λαμβάνω εγώ μια τέτοια απόφαση. Τώρα, οι εμπειρογνώμονε ε, έρχονται και ε, δουλεύω μαζί μα ε, για ορισμένε ημέρε ανάλογα με το είδο τη εργασία που πρέπει να κάνουν και σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών, ναι, την εμπλέκουμε στι εργασίε μα, ε, για παράδειγμα σε, σε ζητήματα που σχετίζονται με το HIV, αλλά και για παράδειγμα σε σχέση με τα νέα σχέδια δράση που είχαμε ω προ τη φυματίωση. Και εκεί ε, υπήρξε συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Επίση, αναφέρθηκα στο ζήτημα ήδη των παρενέργειών του εμβολίου για το τύπο H1N1 ε, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι πως, ε, να επαναλάβω μάλλον, είναι πως οι κλινικές δοκιμές συνεχίζονται, ακόμα θα περάσουν από την κανονική διαδικασία διοδότησης από το EMEA, αλλά αν υπάρχουν συντηριακές παρενέργειες, προφανώς και το ECDC από την πλευρά του θα παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά την κατάσταση. Αναφέρθηκα ήδη στο ζήτημα του εμβολιασμού της γρήπης και απαντώντα σε εσά και πάλι Πρόεδρε, ναι, το κάθε κράτο μέλο έχει το δικό του σχέδιο δράση και δεν έχουν την ίδια ποιότητα αυτά τα σχέδια δράση, αλλά υπάρχει ένα ελάχιστο κοινό πρότυπο γιατί είχαμε μια κοινή, ε, κοινέ κατευθυντήρε γραμμέ ε, από κοινού από τη δική μα πλευρά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, εκπόνηση αυτών των σχεδίων δράση και μετά από την εκπόνησή τους ε, ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο ε, από κοινού με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Οργανώσης Υγείας, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσο τα σχέδια δράσης καλύπτουν ακριβώς τα ίδια θέματα, τα ίδια προβλήματα, για να ε, κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση και θεωρώ προσωματικά από το 2005 αυτά τα σχέδια δράση έχουν βελτιωθεί πολύ ποιοτικά. Δεν είναι ακόμα όλα ε, στο ίδιο επίπεδο ποιότητας, αλλά είναι ε, ε, παρικοί για να ανταποκριθούν στο στόχο τους, στο φάση δηλαδή της πανδημίας. Υπάρχει ακόμα και ε, αυτή ε, το, η διασφάλιση η οποία θα πρέπει να επιτυχάνεται σε ό,τι αφορά τη συνέχεια αυτών των ε, δράσεων μέσα σε αυτά τα σχέδια και εκείνο που επίσης θα κάνουμε είναι μέσα στο φθινόπωρο η αναθεώρηση των σχεδίων δράσης των κρατών μελών με βάση τις νέες πληροφορίες που θα έχουμε λάβει σε ό,τι αφορά το, τη γρήπη. Δηλαδή ακόμα οριστικοποιούνται τα σχέδια ετοιμότητας των κρατών μελών. Νομίζω πως απάντησα σε όλα τα ερωτήματα στο πρώτο γύρο ερωτήσεων, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Ιάκαμ, για αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Κυρία Φρανσουάς Κουστές, ως πρώτη για το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε για όλα αυτά τα επίκαιρα θέματα. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκδώσει μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα της πανδημίας και για την αναγκαιότητα να μην ξεχάσουμε τον ε, κανονικό εμβολιασμό για την εποχιακή γρήπη. Το υπογραμμίσατε και εσείς. Από όσο ξέρουμε, τα κράτη-μέλη στρέφονται περισσότερο στην αξία του θέματος του ε, ρίσκου της πανδημίας του H1N1 και δεν είπαν τίποτε για την ανάγκη να εμβολιαστεί κανείς κατά τη συνήθους γρήπης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ε, κίνδυνος αντιπαράθεσης, διότι πιστεύουν κάποιοι ότι κάποιες χώρες αντιδρούν υπερβολικά, κυρίως πριν να φτάσει πρώτον πυλών η γρήπη και όταν αρχίσουν κάποια θανετηφόρα κρούσματα, πανικοβάλλονται οι πάντες και όλοι απαιτούν να εμβολιαστούν. Αυτό λοιπόν είναι, που είναι επικίνδυνο είναι ότι η υπερβολική δημοσιότητα που δόθηκε για τον ε, εμβολιασμό αυτής της γρήπης μπορεί να είναι αρνητική σε σχέση με ότι θα πρέπει ο να εμβολιάζεται για τη συνήθη γρήπη. Θα πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Λέτε ότι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτώβριου, αλλά πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνουν ε, από επιστημονικής ε, πλευράς κάποιες ανακοινώσεις για να καλυφθούμε για να υπάρξει και εμβολιασμό κατά τη εποχιακή, τη συνήθου γρήπης. Για να μην μα πούνε εκ των υστέρων, ακούστε, εσείς είστε ε, υπέρ των ε, φαρμακοβιομηχανιών που κάνουν αυτό το ειδικό εμβόλιο Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν, ώστε να μπορέσει κανείς να προστατευτεί από την συνήθη γρήπη. Και η υπερβολική διαφήμιση για την H1N1 να μην οδηγήσει σε αρνητική στάση του πληθυσμού κατά τη συνήθους γρήπη. Τώρα, φεύγω από τη γρήπη και θα ήθελα να φέρω κάτι που εσείς ε, αναφέρατε επίσης η αύξηση των κρουσμάτων φυματίωσης. Πιστεύουμε ότι έχει εκκριζωθεί η φυματίωση από την Ευρώπη. Σήμερα ξαναεμφανίζονται τέτοιου κρούσματα, δυστυχώ, ποιε είναι οι προτάσει που επιβάλλετε εσείς να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λέει ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Γιάκα για την παρουσία της αλλά και για την δουλειά της, διότι πραγματικά τώρα σε τέτοιες στιγμές μπορούμε να εκτιμήσουμε την σημασία ενός οργανισμού λαμβάνοντα υπόψη την δουλειά που κάνει. Και πραγματικά χαίρομαι, είμαι ιδιαίτερα περήφανο που έχουμε ένα τέτοιο οργανισμό, ο οποίο εξυπηρετεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τόσο αποτελεσματικό τρόπο. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για το θέμα που μας απασχολεί, διάβασα κάτι, δεν είμαι πυρογνώμονας εγώ βέβαια, εγώ σε άλλα θέματα είμαι ειδικό Διάβασα μία πρόταση ότι, που λέει ότι σύμφωνα με μαθηματικούς υπολογισμούς μπορούμε να περιορίσουμε την χρήση του εμβολίου και με βάση τις ε, τους, τους, τους υπολογισμούς, με βάση τους υπολογισμούς αυτούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εμβολιασμό μόνο στους φορείς της ασθένειας και όχι μόνο στους αδύνα, στις ε, αδύναμες ομάδες. Καταρχάς, να ρωτήσω αν είναι αλήθεια αυτό που διάβασα. Δεύτερον, ο τρόπος μόλυνσης και διάδοσης αυτών των ε, μικροβίου των νοιών. Είναι μέσω της εισπνοής. Επομένως, οι γενικοί κανόνες υγιεινής και καθαριότητας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Όμως και μια καλή, ένας καλός εξαερισμός των ε, κατοικιών ή των ε, νοσοκομείων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και ίσως θα έπρεπε να προβλέψουμε και έναν και μία μέθοδο ε, χορήγησης των εμβολίων δια της εισπνοής και όχι μόνο μέσω ενέσεων. Και αυτό θα ήταν πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο, διότι με τον τρόπο αυτό το εμβόλιο ή τα φάρμακα τέλο πάντων θα ακολουθήσουν την ίδια οδό που, θα, που ακολουθεί και ο ιός. Και ρωτώ, Πώς σας φαίνεται αυτό. Ε, το κέντρο σας έχει εκτιμήσει, έχει αξιολογήσει, έχει μελετήσει αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιάκοβ για την παρουσία της στην Επιτροπή. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Ε, αυτές τις μέρες, τουλάχιστον στην Νότια Ευρώπη, ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γιάκοβ τι προτείνει το ECDC ακριβώς για τα σχολεία και για την ε, πρόληψη της πανδημίας ε, στον ευαίσθητο αυτοπληθυσμό. Ευχαριστούμε την κυρία Ιάκοβ για την παρέμβασή της. Τον τελευταίο καιρό Βλέποντας ποιες είναι οι πληροφορίες που έδωσαν τη διάφορα κάτι, θα μπορούσα να πω ότι φαίνεται ότι υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια. Σήμερα είπανε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι οι έγκυος, οι μεγάλοι, τα νέα παιδιά. Φαίνεται όμως σήμερα να ακούω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να δούμε πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι πολίτες και μετά να εμβολιαστούν οι έγκυες γυναίκες και, οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά. Από το 2005 πρέπει να πω ότι υπάρχει στα κράτη-μέλη ένα ε, καλό σύστημα πληροφόρησης προς εσάς. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι λαμβάνοντα υπόψη κάποια κριτήρια γενικά για να οριστούν οι ευάλωτε ομάδες είναι η εξή. Μπορούμε να πούμε ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμό σε αυτό το τομέα λειτουργεί σωστά και όλες οι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια εντοπισμού των ευάλωτων ομάδων και τα ίδια μέτρα, κυρίω όσον αφορά την διάδοση τη σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ο Thank you, Mr. President. And... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιάκομπς για την εξαιρετική παρουσίασή της. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, όπως είπατε, προσπαθούμε από τον περιορισμό να φτάσουμε στη μετρίαση, στην άμβλιαση. Πώς αξιολογείτε τη σχετική προσπάθεια για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια μαθήματα πρέπει να αποκομίσουμε κυρίως σε περίπτωση που θα έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την γρήπη ή κάποια άλλη πιο παθογεν, κάποιο άλλο πιο παθογενές νόσημα. Σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβάνεις της δικής μου, έχετε μελετήσει τη αύξηση κάποιων ε, τέτοιου είδους μεταδοτικών ασθενειών. Κύριε Πρόεδρε. Ίσως εγώ δεν βρίσκομαι στο ίδιο μήκο κύματο με τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο εδώ και μίλησαν για πανικό. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ ανησυχώ παρά το γεγονός ότι εμπιστεύουμε τη χώρα μου. Μας είπατε κάτι όμως εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει η κυβέρνησή μας. Διερωτώμε. Πρέπει να πιστεύουμε αυτά τα οποία μας λέει η κυβέρνηση στη Σουηδία Δηλαδή ότι θα πρέπει όλοι να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε στι αρχέ Οκτωβρίου. Είπε η κυβέρνησή μα ότι θα πρέπει να αρχίσουμε πρώτα από τι έγκυε, από τα παιδιά, από αυτού που πάσουν από κάποια χρόνια πάθηση και γύρω στα μέσα Νοεμβρίου να σκεφτούμε κι εμεί οι υπόλοιποι που δεν έχουμε πρόβλημα να εμβολιαστούμε. Εμεί μα είπατε όμω ότι δεν θα υπάρξει εμβολιασμό για τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μας λέτε κάτι διαφορετικό, πράγμα το οποίο γενικά μπορεί να προκαλέσει ανησυχία. Αυτό το οποίο εμένα επίσης με απασχολεί είναι ότι στη χώρα μου τα σχολεία άνοιξαν εδώ και τρεις εβδομάδες. Το δικό μου το παιδί α, πήγε στον Ήπιο και τίποτα δεν έχει προβλεφθεί μέχρι τώρα ε, στα σχολεία για την προστασία των παιδιών και των δασκάλων βεβαίως. Στην Σουηδία επεκτάθηκε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα η γρήπη αυτή. Πώς μπορεί να ενημερωθεί κανείς ε, σωστά και πώς μπορεί να λάβει γνώση όλων αυτών των στοιχείων μας παρουσιάσατε εσείς σήμερα. Κάποιος συνάδελφος επίσης το θέμα της επανεμφάνισης κρουσμάτων φυματίωσης. Όλα αυτά έχουν σχέση με το ρόλο που πρέπει να παίξει κάθε κυβέρνηση και την ανθεκτικότητα του καθενός μας στα διάφορα αντιβιωτικά. Διότι γίνεται λόγος εδώ για ανθεκτικότητα των ζώων στην αντιβιωτικά. Διαρωτώ αν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ όλων αυτών των οποίων λέγονται και των ε, εμβολιασμό. Ασχοληθήκατε με αυτά τα θέματα. Έχετε κάνει κάποιες στατιστικές. Τι έχετε να μου πείτε για αυτό το θέμα συγκεκριμένο. Επιτρέψτε μου και εμένα να θέσω κάνα δύο ερωτήματα. Ε, γιατί ε, μας απευθύνονται ερωτήματα τόσο από τους πολίτες μας όσο και από τα μέσα ενημέρωσης. Ε, μας λέτε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι περιοχή του κόσμου. Ε, Ποιο ήταν ο συντονισμό που έγινε μεταξύ των κρατών μελών, ε, των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε πω υπάρχουν κάποια ελάχιστα πρότυπα για τα σχέδια δράση των κρατών μελών. Υπήρξαν κάποια ελάχιστα πρότυπα και για την ε, πρόληψη. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ε, συστάσεις ε, στη Γερμανία για παράδειγμα ε, ε, τα οποία κάποια μέτρα εφαρμόστηκαν από κοινού, κάποια όχι. Για παράδειγμα στην πρώτη μέρα που πήγαν στο σχολείο τα παιδιά έπρεπε να μάθουν πώς να πλένουν με το σωστό τρόπο τα χέρια τους και να το κάνουν συχνά και ούτω καθεξής. Επίσης άλλο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη. Ακούω ότι θα πρέπει οι σταθμοί οι μονάδες ε, εντατική ε, παρακολούθησης των ασθενών ε, θα πρέπει να διπλασιαστούν. Δηλαδή λέτε ότι αν ένα νοσοκομείο έχει 20 κλίνες σε αυτές τις μονάδες θα πρέπει να τις κάνει 40. Είναι κάτι τέτοιο δυνατό από τεχνική άποψης. Επίσης, τέθηκε και το εξή ερώτημα. εάν πει ένα κράτος μέλος πολύ απλά δεν δύναμε, δεν μπορώ. Τι θα το πούμε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, απλά θα το πούμε ατυχήσατε και θα χρειαστεί να ε, βιώσετε έναν υψηλό, υψηλότερο αριθμό κρούσματων. Αυτές λοιπόν οι τελευταίες ερωτήσεις από την προγράμμα μου έχετε τώρα το λόγο. Θα αρχίσω κύριε Πρόεδρε με το τελευταίο θέμα το οποίο θίξατε κι εσείς για τον συντονισμό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ε, ε, ΕΚΠΕ και στις Εθνικές Αρχές, με βάση οι μεθόδους και συστήματα οι μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε τις προεδρίες οι οποίες και κυρίως η Σουδική Προεδρία η τελευταία που ηγούνται αν θέλετε ε, των, της, εφαρμογής των συστημάτων αυτά, αυτών και ο Επιτροπός ο κ. Χιπριανού πριν και η κυρία Βασιλείου τώρα ε, επιβλέπουν τα πράγματα. Έχουν γίνει επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις όπου συζητώνται τα θέματα αυτά και η Σουηδική Προεδρία ξεκίνησε ένα ε, workshop για την πανδημία, θα υπάρξει και ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών και μετά θα υπάρξει και μια ανακοίνωση της ε, Κομισιόν για την πανδημία και για τα θέματα εμβολιασμού. Εκεί θα θυχθούν και θέματα όπως πρέπει να το θέματα της αλληλεγγύης και θα δούμε και τα αποτελέσματα της ε, άτυπης συνόδου των Υπουργών. Ε, υπάρχουν ε, ε συμφωνίες ανάμεσα σε κάποιες χώρες. Άλλες χώρες όμως δεν, είναι, δεν έχουν αυτό το σχέδιο προετοιμασίας για την πανδημία και για την αγορά των εμβολίων. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα κυκλοφορήσει το εμβόλιο αυτό στην αγορά τους. Αυτά είναι θέματα τα οποία ζητήθηκαν και στο τελευταίο Συμβούλιο και θα υπάρξουν και εξελίξεις. Επίσης να σας πω ότι ε, στις, ε, στα πρώτα στάδια αυτής της πανδημίας ε, είχαμε από την αρχή μια τηλεδιάσκεψη αν θέλετε κάθε μέρα εμείς, ε, η Ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα και τα κράτη-μέλη. Και υποβάλαμε εμείς ε, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας ε, για να τα υποβάλαμε στην Κομισιόν για σχολιασμό και για την περαιτέρω επεξεργασία και διαχείρισή τους. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά ανήκαν στα κράτη-μέλη και αυτό θέλαμε να το τονίσουμε η συνεργασία αυτή ανάμεσα στο ΕΚΠΕ στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, εμείς ε, λειτουργούμε σαν διαχειριστές, αν θέλετε, σαν διευθύνοντες όσον αφορά την υποβολή των επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων. Εμείς ε, έχουμε, ε, αν τα, την επιστημονική, προσφέρουμε την επιστημονική υποστήριξη. Υπάρχει μια τριμερή συνεργασία, επομένως, ε, η οποία πρέπει να λειτουργεί σωστά και χαίρομαι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι υπάρχει αυτή η, η, η αγαστή τριμερή συνεργασία εδώ και χρόνια και νομίζω ότι κυρίως στην, στα πλαίσια της πανδημίας αποφελήθηκαμε ιδιαίτερα. Να σας πω επίσης ότι Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και ε, που, αφορούν τα, και που αφορά τον εμβολιασμό για την εποχιακή γρήπη. Βλέπουμε και τον κατάλογο, ανάλογα με, την, ε, με τα κρούσματα, ε, βλέπουμε για τις, ποιες είναι οι χώρες που ανήκουν τον κατάλογο των χωρών που απαιτείται εμβολιασμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο και από την εποχιακή γρήπη πεθαίνουν χιλιάδες, πεθαίνουν χιλιάδες στην Ευρώπη, άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα εμβόλια είναι στη διάθεση των ε, πολιτών. Και αυτό το λέω κάθε φορά όταν συναντιόμαστε με υπουργούς, ε, θα πρέπει να ε, ξέρουμε πόσα εμβόλια έχουν, πρέπει να ξέρουν ε, πόσα εμβόλια έχουν και πόσα χρειάζονται για να καλύψουν ε, τις ε, ανάγκες τους. Και εδώ νομίζω ότι και η Επιτροπή σας μπορεί να βοηθήσει, διότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να επαναλαμβάνονται συνέχεια. Για την φυματίωση τώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό τη, τα κρούσματα φυματίωσης μειώνονται. Όμως το πρόβλημα ποιο είναι ότι στα κράτη, τα νέα κράτη-μέλη που, προ, που προσχώρησαν το 2004 είχαν ε, μεγάλο αριθμό κρουσμάτων φυματίωσης. Τα, οι χώρες της Βαλτικής. Ε, έχει βέβαια σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δεν αυξάνονται ο αριθμός των κρουσμάτων. παρόλα αυτά η κατάσταση κρίνεται σοβαρή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε να προετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, κατά της φυματίωσης. Το κάναμε, ε, υιοθετήθηκε μέσα στα πλαίσια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Τώρα περνάμε στη φάση εφαρμογής και υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη με τα εθνικά τους προγράμματα για να ε, μειωθεί η φυματίωση, να περιοριστεί η φυματίωση. Επίσης, για τη Σουηδία. Ε, να σας πω ότι ε, μία από τις προτεραιότητές μας ε, είναι η χρήση των αντιβιωτικών από τους ανθρώπους όμως. Ε, εμείς ασχολούμεθα με τους ανθρώπους και όχι τόσο με τα ζώα. Άλλος είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνο για την χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα και ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπάρχουν πολλά στοιχεία που αφορούν ε, την χρήση των αντιβιωτικών από τους ανθρώπους. Και τώρα θα πρέπει να δούμε στα διάφορα κράτη πώς εφαρμόζονται αυτά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού, του, Ευρωπαϊκού, του Συμβουλίου γενικότερα. Γιατί ε, θα πρέπει να δούμε πόσο ελεύθερα χορηγούνται τα αντιβιωτικά και πολλούνται τα τα βιβλιοτικά ε, στις διάφορες χώρες, με συνταγή ή χωρίς συνταγή. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα ε, στην Σοβορά και στο Νότο. Στις βόρειες ε, χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο να, έχει, να, να αγοράσει αντιβιωτικά, διότι χρειάζεσαι συνταγή συγκεκριμένη από τον γιατρό. Και πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη η χρήση των αντιβιωτικών για να μπορέσει να τα αγοράσει. στο Νότο τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά και υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά που βλέπετε ανάμεσα στο βορρά και στο νότο ε, και από εκεί ξεκινάει και η, αντίσταση των ε, μικροβίων, των ε, διαφόρων ιών στα αντιβιωτικά. Ε, γιατί η μεγάλη χρήση αντιβιωτικών κάνει τους ιούς να ανθίστανται στη χρήση των, ε, των αντιβιωτικών. Και υπάρχει ε, και μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που είναι η στη χρήση, Ευρωπαϊκή Μέρα για την ευαισθητοποίηση στα αντιβιωτικά, όπου ακριβώς ενημερώνουμε το κοινό για την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών. Ε, τώρα να απαντήσω στον Πίτερ Λίζε για την ε, κλιματολογική αλλαγή, ξέχασα να το κάνω αυτό πριν. Αυτό το οποίο προτιθέμεθα να κάνουμε είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές τράπεζες δεδομένων στις διάφορες επιτροπές ε, και στους οργανισμούς των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετερολογία, ε, ε, ε, για μετεωρολογικά θέματα, τράπεζα δεδομένων για το περιβάλλον, για την τράπεζα δεδομένων για, τις, για τη διάδοση των ασθενειών κτλ. Αυτές οι τράπεζες δεδομένων δεν είναι συνδεδεμένε μεταξύ τους. Αν βρούμε έναν τρόπο να, συνδυάσουμε και να συνδέσουμε τις τράπεζες αυτές δεδομένων, πιστεύω ότι θα υποφεληθούμε περισσότερο από αυτή την συντονισμένη, συνδυασμένη γνώση και θα μπορέσουμε να ε, εξετάσουμε και την αλλαγή του κλίματος και, τις, ε, και τη μετάδοση των διαφόρων ασθενειών. Τώρα βέβαια είμαστε σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Τώρα, ερώτηση του κύριου Πρόντι για τις εισπνοές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, από την εισπνοή είναι ο ένας ε, τρόπος ε, διάδοσης της νόσου, ο άλλος είναι από τα χέρια. Γι' αυτό είπαμε να τα πλένουμε. Δεν το έχουμε εξετάσει αυτό που είπατε εσείς, ε. αλλά θα το λάβουμε υπόψη μας, διότι ας στα, αεροπλάνα, μέσω του συστήματος εξαιρισμού μπορεί να μεταδοθούν μολυσματικές ασθένειες ή παραδείγματος χάρη σε διάφορα σπίτια με τον κλιματισμό κτλ. Όντως, η πρότασή σας ε, είναι πολύ σημαντική. Θα, το, θα την μελετήσω και σας ευχαριστώ που το θίξετε. Τώρα, για το κατά πόσο θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Πολύ καλό το ερώτημα σας, το έχουμε συζητήσει. Εμείς δεν λέμε να κλείσουν τα σχολεία. Όμως, Μπορεί να αναγκαστούμε να κλείσουμε τα σχολεία εάν ας πούμε αρρωστήσουν οι δάσκαλοι, αρρωστήσουν οι μισή, τα μισά παιδιά. Εκεί όντως θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το, το σχολείο. θα πρέπει για να κλείσουμε ένα σχολείο θα πρέπει να σταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα με τα μειονεκτήματα. Ε, τι, ε, πόσο θα διαταραχθεί η, η, η κοινωνική ζωή. Ε, γιατί εάν κλείσει το σχολείο θα πρέπει να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Δεν μπορεί να τα, τα στέλνει στην παιδική χαρά. Το πρόβλημα είναι εάν μείνουν στο σπίτι ποιο θα τα κρατάει. Οι γονεί. Εάν μείνουν οι γονεί δεν θα υπάρχουν υπηρεσίε. Ε, θα πρέπει να περιοριστούν δηλαδή οι βασικέ υπηρεσίε ε, που προσφέρουν στου πολίτε σου. Ε, επομένως θα πρέπει όλα αυτά να τα σταθμίσουμε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, όταν φτάσουμε στην, στο ζενήθ, αν θέλετε, τη ε, πανδημία, ενδεχόμενα θα πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά στο σπίτι. Αλλά τέλο πάντων, θα πρέπει να το σταθμίσουμε. Στην Αμερική, ε, το, στην Ατλάντα, το συζητάνε, αποφασίσανε, μετά από συζήτηση, ενδελεχή συζήτηση, αποφασίσανε να μην κλείσουν τα σχολεία. Στην Ευρώπη το συζητάνε ακόμα. Εμείς όμως δεν συνηγορούμε, δεν λέμε να κλείσουν τα σχολεία εκ των προτέρων. Εκτός και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και τότε αναγκαστούμε να το, να το κλείσουμε. Γιατί στο κάτω-κάτω και αν δεν πάνε στο σχολείο τα παιδιά μπορεί να κολλήσουν από κάπου αλλού. Εφόσον διαδοθεί ευρύτερα ο ιός. Τέλος πάντων, ακόμα είναι κάτι το το, είναι ένα θέμα το οποίο μελετάμε. Τώρα, νομίζω ότι απήντησα και για τα θέματα συντονισμού. Πηγαίνει, είναι πολύ καλό ο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τώρα, οι στρατηγικές περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι ε, ήταν πολύ θετικές θετικά τα μέτρα και οι στρατηγικές ε, Είδαμε πώς συντονίστηκαν οι πολιτικές αυτές ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, νομίζω ότι εξέτασαν την επιδημιολογική κατάσταση πολύ προσεκτικά τα κράτη-μέλη για να περάσουν από το ένα στάδιο, το στο στάδιο περιορισμού, στο επόμενο στάδιο. Τώρα βέβαια έχουμε και την εμπειρία από τα διάφορα στάδια της εξέλιξης της πανδημίας και νομίζω ότι οι μελλοντικέ γενιές θα ε, εξάγουν τα συμπεράσματά του όσον αφορά την πολιτική συγκράτηση. Τώρα, για την παράνομη μετανάστευση. Αυτό είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως το συζήτησε και η Πορτογαλική Προεδρία. Έχουμε συντάξει ένα έγγραφο για, το συνέπεια, για τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης ε, στην, ε, ε, στην διάδοση ασθεν, ασθενειών, όπως είναι παραδείγματο χάρη οι μαγουλάδες, οι παροτίτιδα τέλο πάντων, οι ε, η φυματίωση. Ε, αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Τώρα, στο συνάδελφο από τη Σουηδία να πω ότι έτσι όπως σας είπα οι κλινικές δοκιμές ακόμα συνεχίζονται για, για το εμβόλιο για την νέα γρήπη και εξαρτάται τώρα πότε θα ολοκληρωθούν οι κλινικές δοκιμές, για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν οι κλινικές δοκιμές. Μετά θα υπάρχει μια ταχύτατη διαδικασία ε, εγγραφής, καταχώρησης και έγκρισης. Εάν επομένως οι κλινικές δοκιμές είναι θετικές και ολοκληρωθούν εγκαίρως, εάν ολοκληρωθεί και η γρήγορη διαδικασία, και αν ε, τα, οι ενδείξεις που θα έχουμε από τις κλινικές δοκιμές ε, συνηγορούν ε, πιστικά για την χρήση του εμβολίου, εμβολίου θα δούμε το φθινόπωρο κάποια στιγμή τον Οκτώβριο-Νοέμβρη να κυκλοφορήσουν τα πρώτα εμβόλια. Προφανώς στο πρώτο στάδιο δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλους τους ενδιαφερομένους, διότι η παραγωγή χρειάζεται κάποιο χρόνο και θα συνεχίσει η παραγωγή του εμβολίου μέχρι ότου καλυφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό θα γίνεται σταδιακά. Εάν όμως όλα πάνε ε, βάση του προγράμματος, μέχρι το τέλο Οκτωβρίου, τα, οι πρώτες ε, παρτίδε των εμβολίων θα κυκλοφορήσουν στην αγορά όχι για τις ομάδες κινδύνου. Για τις ομάδες κινδύνου, από όσο ξέρω, οι, οι κλινικές δοκιμές συνεχίζονται. Θα συνεχιστούν και μετά. Αν θα ξεκινήσουν μετά για τις έγκυες και τα παιδιά. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα απευθυνθούμε μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ε, σε εσάς. Ε, διαπιστώνουμε τώρα πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του ECDC και βέβαια θα πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς γρήγορα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη συμμετοχή μας στην στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC. Η συνεδρία Σύλληξη, Ευχαριστώ και του Ερμηνείς ο Πρόεδρος. Και αύριο συνεχίζουμε και στι 10.30, 9 η ώρα συνεδρία των συντονιστών.